lovers. Eva. Allora, we can. Prego, vi chiedo di prendere i posti. Παρακαλώ καθίστε. Sit down, please. Thank you to be here. Grazie di questa... Σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Η συνεδρίαση των συντονιστών ε, καθυστέρησε κάπως. Όπως βλέπετε δεξιά μου έχουμε μια προσκεκλημένη, την κυρία Ντόρις Πακ, που ήδη ήταν παρούσα σε αυτή την επιτροπή και τώρα έχει αναλάβει το ρόλο του συντονισμού για το βραβείο Λούξ. Σε λίγο θα της δώσουμε το λόγο για να μας αναφέρει τις ε, προοπτικές της νέας έκδοσης του βραβείου Λούξ. Ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κινηματογραφικό βραβείο έχει δημιουργηθεί από το Κοινοβούλιο και εμείς ε, του προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Τα τη συνεδρίαση να σας ενημερώσω ότι η συνεδρία στο συντονιστό συζήτησε σχεδόν όλα τα θέματα στην ημερησία διάταξη. Όμως ζητήσαμε να αναβάλουμε ένα σημείο για να οργανώσουμε την ημερησία μας διάταξη και θα συζητήσουμε ένα θέμα που αναβλήθηκε την επόμενη φορά. Τώρα πρέπει να περάσουμε στην έγκριση της ημερησίας διάταξης για να μπορούμε κατόπιν να εγκρίνουμε και τις συστάσεις των συντονιστών. Όπως σας είπα, αυτό θα το αναβάλουμε μετά την ανταλλαγή ε, απόψεων για το σινεμά στην ψηφιακή εποχή. Συμφωνείτε με αυτή την τροποποίηση με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Πρέπει να εγκρίνουμε, θα τα έχετε διαβάσει βέβαια, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 22ης Ιουλίου και 3-4 Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Εντάξει, και περνάμε στο σημείο 4. Σήμερα θα έχουμε γραμματεία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσέχικα, στονικά, ουγγρικά, πολεμικά, βουλγαρικά και ρουμάνικα. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 11 Νοεμβρίου και όχι στις 10 θα έχουμε μια πολύ σημαντική ακρόαση όπου έχουμε προσκληθεί από την Επιτροπή Γιουρί για την μελλοντική ανάπτυξη του copyright στην Ευρώπη και θα συμπροεδρεύουμε εμείς ε, και όπως ξέρετε είναι συνδεδεμένη η Επιτροπή μας με το θέμα αυτό. Έχει αλλάξει ε, η ημερομηνία, είναι στις 11 Νοεμβρίου από τις 3.30 μέχρι τις 6.30 και έχοντας κατά νου τη δυνατότητα να έχουμε μία ισχυρή συνεργασία με την Επιτροπή Γιούρη, θα παρακαλούσα όλα τα μέλη της δικής μας Επιτροπής να είναι παρόντα σε εκείνη την ακρόαση. Και τώρα... Να περάσουμε στο θέμα για το οποίο έχουμε καλέσει εδώ την κυρία Πακ. Ξέρετε ότι έχει ασχοληθεί με το βραβείο Λούξ από την αρχή, από τη γέννησή του. Ξέρετε το ρόλο που έχει διαδραματίσει στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και εγώ αυτά τα πέντε τελευταία χρόνια έχω παρακολουθήσει εκ του σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε μεταβεί και σε κάποια φεστιβάλ της Βελετίας, του Κλουβιβάρη και θεωρήθηκε αυτό το βραβείο ως μια ευκαιρία για να ε, προωθήσουμε τους ε, νέους Ευρωπαίους κινηματογραφιστές ε, για θέματα ευαίσθητα για την Ευρώπη και είχαμε μια συμμετοχή πολλών χωρών σε αυτό το διαγωνισμό, το Λουξ μεταξύ άλλων. Γνωρίζετε ότι μετά την πρώτη επιλογή των πρώτων 10, τελικά όλοι οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή της ε, ταινίας που θα κερδίσει το βραβείο. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εσείς ε, να τοποθετηθείτε επί των τριών νέων κινηματογραφιστών. Πρόκειται για τρεις ταινίες ε, μεγάλης ποιότητας έχουν ήδη παρουσιαστεί αυτούς τους μήνες σε κάποια σημαντικά σε κάποιες σημαντικές κινηματογραφικές εκδηλώσεις. Επίσης, ε, μεταφράζεται η ταινία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο υποτιτλισμός αποτελεί μία από τις δράσεις του προγράμματος Μέντια της Δημιουργικής Ευρώπης. Είναι σημαντικό κυρία Πακ και επειδή έχει δεσμευτεί τα μάλα κατά τη γένεση του βραβείου και την πρόθεσή του, της ανέθεσε ο πρόεδρος Σούλτς ε, τη θέση της συντονίστριας για το βραβείο. Εγώ θα ήθελα να διαβεβαιώσω την Τόρις ε, ότι εμείς θα συνεχίσουμε ως Επιτροπή Πολιτισμού να δεσμευόμαστε για την προώθηση του βραβείου αυτού. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε και την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ Σίλβια. Καλημέρα, θα μιλήσω γερμανικά. δεν μιλώ επαρκώς Ιταλικά. Ε, Ευχαριστώ την Πρόεδρο και τη Γραμματεία και τους συντονιστές για το γεγονός ότι έχω την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα. Το Προεδρείο του Κοινοβούλιο την άνοιξη με, ε, ανέδειξε ε, συντονίστρια για αυτό το βραβείο Λουξ. Μάλλον από το φόβο τους ότι σε περίπτωση που το νέο κοινοβούλιο δεν είχε ενδιαφέρον ε, για αυτό το βραβείο, θα χρειαζόμασταν κάποιον ο οποίος δεν θα ήταν πλέον βουλευτής μετά από 25 χρόνια ε, ως ευρωβουλευτής. Εγκατέλειψα το κοινοβούλιο και αφιερώνω τη ζωή μου πλέον στον πολιτισμό και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ γιατί μπορώ να σας μεταδώσω κάτι από τη φλόγα που καίει μέσα μου για, αυτήν την, ε, για αυτό το βραβείο. Δεν θυμάστε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά πριν από 10 χρόνια ο Βιμ Βέντερς εκφώνησε μια μεγάλη ομιλία, μια πολύ σημαντική ομιλία στο Βερολίνο και είπε ότι σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης, σε αυτούς τους καιρούς όπου πολλοί άνθρωποι στρέφουν την πλάτη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, θα πρέπει να βρούμε δυνατότητες να αναζωογονήσουμε το ευρωπαϊκό όνειρο. Και γι' αυτό θα πρέπει να διηγηθούμε ευρωπαϊκές ιστορίες. Ευρωπαϊκές ιστορίες σημαίνει ευρωπαϊκές ταινίες, προβολή ευρωπαϊκών ταινιών. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Δημιουργήσαμε αυτό το βραβείο τότε, ήταν το τμήμα επικοινωνίας του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με την Επιτροπή εδώ. Δημιουργήσαμε αυτό το βραβείο για να αξιοποιήσουμε με ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες να δημιουργήσουμε γερμανικές, εστονικές, σλοβενικές ταινίε και ώστε αυτές να προβάλλονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέραν αυτής. Δεν ήταν εύκολο καθήκον γιατί μας χαρακτηρίζει η πολυγλωσσία. Έχουμε 24 γλώσσες και είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα βραβείο μέσω του οποίου θα υποτιτλίζονται όλες οι ταινίες που συμμετέχουν στον, στο διαγωνιστικό κομμάτι σε 24 γλώσσες. Νομίζω ότι είναι ένα εκπληκτικό βραβείο και νομίζω ότι βοηθά ιδιαίτερα τους μικρούς και τους μεσαίους ε, κινηματογραφιστές και τις ε, εταιρείες διανομής να διανέμουν ε, αυτήν την, τις ταινίες αυτές σε μεγαλύτερο κοινό. Δημιουργήσαμε λοιπόν μια κριτική επιτροπή που κάθε χρόνο ήταν λίγο διαφορετική. Μια κριτική επιτροπή από εξωτερικούς συνεργάτες, από κριτικούς κινηματογράφου, από ακαδημαϊκούς, από ανθρώπους του, του κλάδου που νομίζω ότι ε, συναντιούνται τρεις φορές το χρόνο, την Άνοιξη και από τον τεράστιο θησαυρό ταινιών που προβλήθηκαν την προηγούμενη χρονιά στις αίθουσες κινηματογράφου προσπαθούν από αυτή την, από αυτή την τεράστια ποικιλία όπως είπα να διαλέξουν 10 ταινίες. Αυτές οι 10 ταινίες ε, στη συνέχεια ε, από τις 10 αυτές επιλέγονται 3 που από τις οποίες εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο μετά πρέπει να επιλέξουμε. Στην αρχή υποτιτλίζαμε μόνο την, ε, την νικήτρια ταινία. Το αλλάξαμε αυτό όμως στην, ε, στην ε, πορεία. Από, από την επιλογή των από τη στιγμή της επιλογής των τριών ταινιών υποτιτλίζονται και οι τρεις αυτές στις 24 γλώσσες ώστε να έχει ο καθένας τη δυνατότητα έγκαιρα να δει τις ταινίες αυτές. Έχετε μπροστά σας ένα πακέτο στη γλώσσα σας, όλοι σας. Είναι πολύτιμο, μην το πετάξετε, μην το αφήσετε εδώ. Είναι στη γλώσσα σας, μεταφρασμένο και εκεί θα δείτε και τις ε, τρεις ταινίες υποτιτλισμένες στη γλώσσα σας και εκεί μπορείτε να δείτε και όλη την πορεία και τους στόχους που επιδιώκουμε όλα γραπτός εκεί μέσα. Οπότε εγώ θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις μόνο. Λοιπόν, υποτιτλήσαμε αυτές τις τρεις ταινίε και θα αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι ο νικητής. Λοιπόν, τι θα, τι θα, τι θα λάβει ο νικητής. Ο νικητής θα πάρει και μία έκδοση για τυφλούς ανθρώπους και αυτό είναι κάτι που, που έλειπε πρέπει να σας πω. Η πρώτη ταινία που οργανώσαμε προκειμένου να ε, μπορεί να την παρακολουθήσει ε, και ένας τυφλός, ακούει κανείς τη γλώσσα αλλά ακούει και έναν αφηγητή που εξηγεί στον ε, τυφλό θεατή, ακροατή τι συμβαίνει. Στο Βερολίνο λοιπόν είχαμε συζητήσει με οργανώσεις τυφλών και οι άνθρωποι αυτοί μας είπαν ότι είναι πραγματικά καταπληκτικό και σας παρακαλώ κυρία Πακ κάντε κάτι για να μπορούμε και εμείς να δούμε εντός εισαγωγικών περισσότερες ταινίες. Μας συγκίνησε πάρα πολύ αυτό και γι' αυτό ε, διασφαλίσαμε ότι και οι τρεις ταινίες υποτιτλίζονται έγκαιρα και ο νικητής, ε, η νικήτρια ταινία μάλλον βγαίνει και σε έκδοση για τυφλούς. Και έτσι όλες οι ταινίες αυτές ε, διανέμονται και προβάλλονται και έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες προβολής. Συνεργαζόμαστε με το Άρτε, το δίκτυο Άρτε, που φέτος από τις 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας, στις 8 Ιουνίου, πρόβαλε το, το, το, το Άρτε την ταινία η Ξένη» για τρεις μήνες. Ήταν ε, δωρεάν στην υπηρεσία κατά παραγγελία που, που προσφέρει, που ήταν ταινία που είχαμε βραβεύσει εμείς. Ε, και αυτό είναι φοβερό, διότι... Ε, το Άρτε κανονικά δίνει, ε, προβάλλει ε, περιεχόμενο μόνο στα γερμανικά και στα γαλλικά, αλλά λόγω του ότι υπήρχε αυτή η ταινία, κατάφερε και προβλήθηκε η ταινία αυτή σε ακόμα μεγαλύτερα κενά. Κοινά. Το βραβείο Λούξ αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο πλέον, ακόμα και σε σχολεία. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου προσπαθούν, καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να φτάσει αυτό το ε, βραβείο και στα σχολεία. Ποιο, είναι λοιπόν το θέμα του βραβείου. Εμείς δεν ψάχνουμε ταινία που θα ασχολείται με αυτό το πρόβλημα και θα προτείνει αυτή τη λύση. Εμεί δεν κάνουμε τίποτα. Αυτά έτσι και τα κάνει η Κριτική Επιτροπή. Αλλά γνωρίζετε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο, έχει τέτοια ποικιλομορφία, έχει τόσα θετικά αλλά και τόσα προβλήματα που ε, μπορεί κανεί να τα δει στο Ελσίνκι και στο Παρίσι και στην Αθήνα. Γι' αυτό το λόγο το περιεχόμενο των ταινιών αυτών είναι πάντοτε περιεχόμενο το οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει με τους ανθρώπους που παρακολουθούν την εκάστοτε ταινία. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε και τις ε, ημέρες κινηματογράφου Lux, Lux Film Days. Ε, διοργανώθηκαν τέτοιες εκδηλώσεις ε, στην, σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη. Και είναι κάτι που συγκινεί τους ανθρώπους πραγματικά αν πάτε εκεί, και αυτό είναι, αυτό είναι, και, αυτός, αυτός είναι και ο, ο λόγος που τις διοργανώνουμε. Για εμάς, ως, για σας ως συναδέλφους, γι' αυτό τη δημιουργήσαμε αυτή την εκδήλωση. Για να μπορείτε να συζητήσετε με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τις ταινίε αυτές, για να μπορείτε να, να, να, μιλήσετε για το περιεχόμενο των ταινιών αυτών, για τα συμπεράσματα ε, που μπορείτε να εξαγάγετε κι εσείς για τη δική σας νομοθετική εργασία. Πάρτε για παράδειγμα την ταινία Welcome Νομίζω πριν από δύο χρόνια. Ήταν η ταινία που νίκησε πριν από δύο χρόνια. Ήταν του Λίου Βε. Και έδειχνε πως ένα αγόρι από το Αφγανιστάν κατάφερε να φτάσει με πάρα πολλά προβλήματα βεβαίως στο Καλέ και από εκεί θέλει να πάει στο Ντόβερ της Βρετανίας. Ήταν μια ταινία που ήταν ιδιαίτερα συγκινητική που έδειχνε τα προβλήματα και τι δυνατότητες θα είχε κανείς να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο και είναι ένα πρόβλημα αυτό των, των, ανθρώπων που αναζητούν άσυλο. Εμείς πολλές φορές θα, έλεγα ότι ζούμε σε παραδείσιες καταστάσεις. Δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε τι τραβάνε οι άνθρωποι που ψάχνουν άσυλο. Και η ταινία αυτή είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που πραγματικά σου δημιουργεί την αίσθηση ότι πρέπει, πρέπει να βοηθήσω κι εγώ. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον μετά και για τους συναδέλφους εδώ, τους ευρωβουλευτές, να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα με τους ε, θεατές, για να μπορέσουμε να, να αξιοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία και στην νομοθετική μας δουλειά. Και αυτό αφορά και άλλες επιτροπές, τους αδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για παράδειγμα. Αυτό θέλω να πω. Όπου λοιπόν γίνονται προβολές αυτών των ταινιών, σας παροτρύνω να πηγαίνετε κι εσείς στις προβολές για να μπορείτε να μιλάτε και με τους ανθρώπους και πιστέψτε με, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έρθουν αν τους στείλετε μια πρόσκληση και πείτε ελάτε γιατί θα σας βγάλω μια ωραία ομιλία για την Ευρώπη, για το ευρώ. Δεν θα έρθουν. Αλλά σε προβολή ταινία είναι πιο πιθανό να έρθουν και έτσι μπορούν να μάθουν περισσότερο την, ε, τη δουλειά του Ευρωκοινοβουλίου. Και αυτό είναι άλλωστε και ο σκοπός της όλη διοργάνωση, γιατί την πληρώνουμε την διοργάνωση από, την, από, το, από το τμήμα ε, επικοινωνίας του Κοινοβουλίου. Δεν βγαίνει από τον γενικό προϋπολογισμό αυτό. 600.000 ευρώ το χρόνο. Υπήρχαν κάποιοι ευρωβουλευτές, παλιότερα τουλάχιστον, που λέγανε ότι μα τι μας νοιάζουν εμάς οι, οι ταινίες, ο κινηματογράφος, ας πάνε να βρουν ε, διανομής μόνοι τους οι εταιρείε παραγωγής. Εγώ μπορώ να σας πω, είναι σημαντικότερο από το να φτιάχνουμε στυλό με το λογότυπο του Ευρωκοινοβουλίου, το να φτιάχνουμε Ταινίε που φτάνουν σε χιλιάδες ανθρώπους. Πιστέψτε με, πραγματικά έχω εμπειρία 7 χρόνων και είμαι ενθουσιασμένη με την, όλη, με την διοργάνωση αυτή. Δεν θα πάμε μόνο στις αίθουσες προβολής, θα πάμε και στα, στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωση για να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτές τις ταινίες. Γι' αυτό θα ήθελα όλοι σας να συμμετέχετε στην ε, διαδικασία αυτή. Σήμερα λοιπόν, 3, χθες δηλαδή, 3 Νοεμβρίου, είδατε, ε, ξεκινάμε το screening, τη διαδικασία της προεπιλογής. Λοιπόν, οι ευρωβουλευτές, έχετε ένα DVD μπροστά σας. Αλλά μπορείτε να δείτε και σε video on demand τις ταινίες αυτές, βίντεο κατά παραγγελία. Έχετε τις οδηγίες, δεν χρειάζεται να υπησέλθω σε λεπτομέρειες. Και υπότιτλους σε 23 ε, γλώσσες. Τα DVD είναι μόνο για του ευρωβουλευτέ. αλλά όποιο που, όποιος, πάρει DVD πρέπει και να ψηφίσει. 222 ψήφισαν ε, πέρσι. Νομίζω δηλαδή ότι έχουμε περιθώρια βελτίωση. Υπάρχουν και νέοι συνάδελφοι που είναι ενθουσιασμένοι με αυτήν την ε, με την διοργάνωση αυτή. Λοιπόν, δεν μπορώ να πάω και σε όλες τι επιτροπές, αλλά πραγματικά εσείς θα έπρεπε να γίνετε, να γίνετε ε, οι αυτού του μηνύματο για το βραβείο Λίξ. Ε, ε, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία στη σημερινή εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται τόσο μεγάλη κριτική να αποδείξουμε ότι προσπαθούμε ε, να συγκινήσουμε ανθρώπους για το ευρωπαϊκό όνειρο όπως το εμπνεύστηκε ο Ρόμπερ Σουμάν. Α, ναι. Από τις 2 ως τις 12 Δεκεμβρίου, στο μεσημεριανό διάλειμμα και, και το βράδυ μετά τη συνεδριάση των Επιτροπών, εδώ στην αίθουσα Μέγιο Ντιμέινιν, μπορείτε σε μια μικρή κινηματογραφική αίθουσα που θα δημιουργηθεί ad hoc για αυτήν την ε, περίοδο, να δείτε τις ταινίες. Θα πάρετε και ένα πρόγραμμα ε, προβολών για να μπορείτε να δείτε τις ταινίες αυτές και σε μεγάλη οθόνη. Νομίζω ότι είναι ε, μια πρωτοβουλία που πραγματικά περιπεί μεγάλη τιμή στο κοινοβούλιο. Έχουμε τρεις ταινίες ε, από φέτος. Ε, μια ταινία από τη Σλοβενία, το θέμα της ε, αφορά πολλά σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το class enemy, ο ταξικός εχθρός, ο, ο καθηγητής όμως που δημιουργεί προβλήματα σε μια τάξη. Νομίζω ότι είναι μια ε, καταπληκτική ταινία. Η δεύτερη ταινία είναι μια γαλλική ταινία της Ελίν Σαμά. Μια ταινία για μια συμμορία κοριτσιών, Brand de Fille, Band de Fille. Επίσης εξαιρετική ταινία και σας τη συνιστώ ε, ανεπιφύλακτη. Και μετά έχουμε μια ταινία, την τρίτη ταινία του Παύλ Παυλικόφσκι, είναι διάσημος ε, κινηματογραφιστής Πολωνός που ζει στην Αγγλία, που έχει λάβει ήδη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ε, μάλλον έχουμε τα ίδια γούστα με την ε, Ακαδημία. Και θέλω να σας πω ότι με συγκίνησε σε αυτή την ταινία. Όταν συζητήσαμε για αυτή την ταινία, κάποιος νέος άνθρωπος είπε, ε, και επειδή ξέρετε είναι ασπρόμαυρη η ταινία αυτή, Τότε μόλις συνειδητοποίησα εγώ ότι η ταινία ήταν ασπρόμαυρη. Εγώ στη διάρκεια της προβολής της ταινία δεν το είχα καταλάβει ότι ήταν ασπρόμαυρη. Είναι μια ταινία που είναι πραγματικά συγκινητική, εκτιλήσεται στην κομμουνιστική Πολωνία. Και έχουμε και τα Lux Film Days, σας είπα πληροφορίες για αυτή την ε, διοργάνωση. Και θέλω να σας πω ότι Τις, τις ταινίες αυτές μπορείτε να τις δείξετε και στις εκλογικές σας περιφέρειες. Στις 17 ε, Δεκεμβρίου θα απονεμηθεί το βραβείο Λούξ από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ε, παρουσία των σκηνοθετών και κάποιων ηθοποιών. Όταν λοιπόν απονεμηθεί το βραβείο αυτό, θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε στη συνέχεια αυτή την ταινία στις, στις πατρίδες, στις χώρες σας για να διοργανώσετε προβολές και να μιλήσετε με νέους ανθρώπους. Σας δίνει μια καταπληκτική ευκαιρία να συζητήσετε με όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ότι βεβαίως ότι δεν είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες ε, της ταινίας. Ε, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη διανομή τη ταινία θέλουν και εκείνοι να βγάλουν κάποια χρήματα, προφανώς. Αλλά έχουμε εδώ στο, στο, στο κοινοβούλιο ε, προϋπολογισμούς κάθε ευρωβουλευτής έχει, μπορεί πιστεύω να δώσει κάποια φορά και 300 ευρώ για να νοικιάσει την ταινία αυτή και να, να κάνει να διοργανώσει μια προβολή. Πραγματικά είναι εκπληκτικέ οι ταινίε αυτέ. Μαριζέλα, μπορεί να σηκωθεί λίγο. Και δίπλο ο Γεντρίς, ο Τσέχος. Είναι οι δύο άνθρωποι που διαχειρίζονται τη διοργάνωση και την απονομή του βραβείου και, τον, και τα φεστιβάλ. Λοιπόν, και τέλο να πω ότι νομίζω ότι μπορούμε να μετεξελίξουμε ακόμα περαιτέρω το, το βραβείο αυτό. Για παράδειγμα, να μην υποτιτλίζουμε μόνο τρει ταινίε, ίσω στο μέλλον να μπορούσαμε να υποτιτλίσουμε και πέντε ταινίε ή στο απότερο μέλλον και τι δέκα ταινίε, να υποτιτλίζονται και οι δέκα ταινίε. Γιατί το θέμα που μα ενδιαφέρει είναι να γίνεται προβολή των ταινιών αυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ταινίε αυτέ επιλέγονται από, από τις 28 χώρε μέλη. Οπότε κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτήν την διοργάνωση. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα, μεγάλα μέσα ε, επικοινωνίας, με τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής. Έχουμε πάντως την δυνατότητα να συνεχίσουμε και να μετεξελίξουμε το βραβείο αυτό ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορώ να φανταστώ ότι το βραβείο αυτό μπορεί κάποια στιγμή να ε, μετεξελιχθεί στο σημαντικότερο βραβείο κινηματογραφικό ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε βεβαίως το European Film Award. Υπάρχει και ένα βραβείο της Κομισιόν, αλλά δεν το ξέρει κανείς αυτό το βραβείο. Εγώ το, ξέρω γιατί ήμουν πάντοτε παρούσα όταν απονεμόταν το βραβείο, αλλά γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Νομίζω όμως ότι αυτό το βραβείο Λουξ πρέπει να το ενισχύσουμε ε, και να έρθουμε και σε συνεννόηση με την Κομισιόν για να το προωθήσουμε ακόμη περισσότερο και νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιε δυνατότητε. Λοιπόν, παρακαλώ να συμμετέχετε κι εσεί. Θέλω να σα παρατρύνω να μεταφέρετε κι εσεί αυτό το μήνυμα. Α, και ξέχασα και κάτι ακόμη. Στα Film Days, στα φεστιβάλ προβολή, Όλοι όσοι συμμετέχουν στις προβολές αυτές μπορούν να ψηφίσουν. Η ψηφοφορία αυτή δεν θα επηρεάσει τον νικητή, αλλά είναι μια δημοσκόπηση, ας πω έτσι, μεταξύ των ε, θεατών. Και πέρσι το κάναμε αυτό. Υπάρχει, δίνει και ένα κίνητρο για να πάει κανείς στην προβολή. Και ακόμη, και κάτι τελευταίο, στο πλαίσιο του βραβείου αυτού, στη Βενετία, όταν παρουσιάζονται αυτές οι τρεις ταινίες, εδώ και τέσσερα χρόνια έχουμε μια ε, συνεργασία με το Venice Days, που είναι μια διοργάνωση στο πλαίσιο του φεστιβάλ Βενετίας, όπου, όπου εργάζεται και ο κύριος Μπαζάντη και η κυρία Καστελίνα που ήταν ε, προκάτοχή μας εδώ σε αυτή την επιτροπή και κάθε χρόνο προσκαλούμε έναν νέο συνεφίλ, κινηματογραφόφιλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, όχι κινηματογραφιστή. Και έρχονται λοιπόν 28 άνθρωποι για μία εβδομάδα στη Βενετία και έχουν εκεί την, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, να μιλήσουν με ηθοποιούς, με σκηνοθέτες, να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπορώ να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν την Ευρώπη με έναν τρόπο ιδιαίτερο, πολύ μοναδικό. Ε, γιατί συνεργάζονται με 27 άλλους ανθρώπους και διατηρούν και τις επαφές τους και στη συνέχεια είχα πάει κάποτε στην Περνινάλε και έρχεται ένα άνθρωπο, ένα νεαρό και μου λέει ε, «Είστε η κυρία Πακ» και μου είπε «Εγώ είμαι ένα από του 27, από την Κροατία ήταν». Δεν, υπήρχε, δεν ήταν ακόμα μέλο η Κροατία, ήταν 27 χώρε τότε. Ξαναλέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί γίνονται φίλοι μέσα, αυτή, μέσα, μέσα αυτής της διαδικασίας, διατηρούν υποφέσεις και νομίζουμε ότι προωθούμε την ευρωπαϊκή ιδέα, βάζουμε στο κέντρο τον, πολιτισμό και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μας υποστηρίξετε όλοι σε αυτή τη διοργάνωση και σας ευχαριστώ ε, πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω και να σας ε, παροτρύνω για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Στην Ιταλία λέμε ότι όταν κάποιος έχει πάθος γίνεται αισθητό. Ευχαριστούμε λοιπόν Ντόρις ε, για το πάθος που δείχνεις και εύχομαι κάθε επιτυχία στο βραβείο Λουξ. Εγώ συντορίζομαι για κάποιου άλλου συναδέλφου εδώ στο Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων η κυρία Τρούπ, ε, αυτή την εμπειρία των Venice Days, αυτών των ημερών στη Βενετία και οι τρεις ταινίες που έχουν επιλεχθεί νομίζω ότι θα παρουσιαστούν στη Βενετία. Αρχίζουν ε, λοιπόν ε, να παρουσιάζονται και στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Εγώ θα ενθάρρυνα τους συναδέλφους να δουν τις ταινίε ε, στη μεγάλη οθόνη, όχι στον υπολογιστή αξίζει το λόγο και υπάρχει αυτή η δυνατότητα 2-12 Δεκεμβρίου να τις δείτε στην αίθουσα Μενόη αλλά να καλέσετε ε, και συναδέλφους από τη χώρα σας να δράξουν αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει κάποιος που να θέλει το λόγο για αυτό το θέμα ήταν όλα σαφέστατα. Ράιαν Πέτρα. Παρακαλώ. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ, Doris Πακ, που είσαι εδώ σήμερα και που πάλι δίνεις μάχη για αυτό το έπαθλο, για αυτό το βραβείο. Ήσουν συνειδήτρια και έδωσες την ιδέα για αυτό το βραβείο ταινία. και είσαι πεπισμένη μαχητής ε, για αυτό το έπαθλο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα λοιπόν που ακριβώς στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό πρέπει να αποσταλεί ότι η Ευρώπη όχι μόνο σε σχέση με τα όσα γίνονται για τις ταινίε. Τα ίδια τα ευρωπαϊκά θέματα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των ταινιών. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι πολλές φορές ε, αυτά τα οποία βλέπουμε για την πραγματικότητα και τον προβληματισμό και τις σκέψεις που εκφράζονται, μόνο αμερικανικά θέματα περνάνε στο κοινό. Και όταν βλέπουμε τέτοιου είδους ταινίε από την Αμερική, που είναι, πώς να το πω, κάθονται στα σαλόνια οι Ευρωπαίοι και πλημμυρίζονται εκεί από αμερικανικές ταινίες και δεν έχει καμιά ευκαιρία η ευρωπαϊκή ταινία και λόγω της γλωσσικής πολυμορφίας που έχουμε και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται για την Ευρώπη. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να προσπαθήσουμε με Ευρωπαί... ευρωπαϊκές ταινίες, ευρωπαίους κινηματογραφιστές να έχουμε μια ευκαιρία που θα τους προσφερθεί και να ξεπεράσουμε το γλωσσικό φραγμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να διευκολύνουμε την υπέρβαση αυτή για τα γλωσσικά θέματα και να υπάρξει μια γεφυροποίηση. Ο υποτιτλισμός είναι κάτι κανονικό σε πολλά κράτη δεν είναι όμως πάντα αυτό το οποίο είναι δεδομένο και όλο και περισσότερο μπορεί να προβληθεί και υπάρχουν πολλές δυνατότητες λοιπόν οι υποτιτλισμοί να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο άνετοι και να μπορεί κανείς να δει το βράδυ μια τέτοια υποτιτλισμένη ταινία. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το βραβείο Λουξ. Σε ευχαριστώ για τις προσπάθειές σου και θέλω να επισημάνω ότι για κανέναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει δικαιολογία να μην συμμετέχει και να μην ε, ε, δώσει, να κάνει προσπάθεια σε αυτό το ε, πλαίσιο. Μπορούμε να δούμε και το βράδυ σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή και όσοι έχουν χρόνο μπορούν να αποφασίσουν να δουν αυτές τις ταινίες. Αξίζει. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογία. Όποιος θέλει μπορεί να το κάνει και να παρακολουθεί και πραγματικά όσοι ενεργά συμμετέχουν στις, ε, στην εκλογή θα πρέπει να αυξήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Για τη δική μου ομάδα μπορώ εγώ να πω ότι όλα θα κάνουμε, ό,τι περνά από το χέρι μας να ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους να δουν αυτές τις ταινίε. και έτσι να υποστηρίξουμε κάπως και εμείς αυτό το οποίο εμείς κάνουμε εδώ σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σημαντικό θέμα η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω των ταινιών με τους συντονιστές συζητήσαμε πιο πριν ποιες μελέτες θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση και υπό το πλαίσιο της, κατεύθυ... ταυτότητας που μπορούμε να εκφράσουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα, νοοτροπία ευρωπαϊκή, πώς αντανακλώνται στις ταινίε οι προβληματισμοί, οι, δομή που, οι δομές που έχουμε Όλα αυτά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Χαίρομαι, στη Γερμανία τουλάχιστον υπάρχουν πολλά όργανα και υπάρχουν και πολλές πληροφορίες, γραφεία για τη διάχυση πληροφοριών για αυτές τις ταινίες. Το Σαββατοκύριακο στην Κολονία για παράδειγμα και στο Βερολίνο έχουμε μια εκδήλωση και σε πολλές άλλες πόλεις που δίνουμε συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία. Κάθε ευρωβουλευτής θα είχε τη δυνατότητα στη χώρα του, στην πατρίδα του να συμμετάσχει σε τέτοιες εκδηλώσεις να μπορέσουν να συζητηθούν τα θέματα των ταινιών με τους πολίτες, να δραχθούμε τις ευκαιρίες που προσφέρεται με αυτό το βραβείο, με αυτό το έπαθλο ταινία να συμμετάσχουν οι πολίτες περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πέτρα και κατόπιν ε, επόμενο συνάδελφο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Doris Πάκα για το ότι όπως ε, συνήθως γνωρίζουμε με μαχητικό τρόπο για τους πολλούς νέους συναδέλφους που είναι μέλη αυτής της Πολιτιστικής Επιτροπής εξοικειώνει τα θέματα για το βραβείο ταινία. Δεν θέλω, δεν έχω να προσθέσω πολλά από τα δικά μου βιώματα να αναφέρω κάποια πράγματα. Από τότε που είμαστε στο Κοινοβούλιο κάθε χρόνο όταν αποδίδεται, δίνεται αυτό το έπαθλο σε ένα μικρό κινηματογράφο στο Düsseldorf δείχνουμε το τι έχει συμβεί και τις ε, ταινίε. Μπορώ να το συστήσω αυτό σε όλους. Μικρές αίθουσες κινηματογραφικές που μπορούν να υποστηριχθούν. Αυτό κάνουμε και στο Düsseldorf. Αποκινούμε μια ε, μικρή τέτοια κινηματογραφική αίθουσα Κάτι κοστίζει, λίγα ευρώ κοστίζει όλα και όλα, αλλά αξίζουν οι ταινίες να τύχουν αυτής της υποδοχής. Και οι πολίτες στους οποίους μπορούμε να φτάσουμε με τέτοιες πρωτοβουλίες, με κανένα άλλο τρόπο δεν θα πήγαιναν σε κάποια άλλη ας το πούμε τέτοια ε, πρωτοβουλία αλλά όταν προσκαλούνται στο βραβείο Λουξ για τις κινηματογραφικές ταινίες και τους λέμε είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία που αντανακλά την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τους ευρωπαϊκούς προβληματισμούς, γεμίζει τότε η αίθουσα και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει ένας σημαντικός εμπλουτισμός διότι κάνουμε κάτι παραπάνω για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ταυτότητα με τέτοιες δράσεις από ότι με πολλές άλλες θεματικές πρωτοβουλίες που όλες τους μπορεί να είναι σημαντικές αλλά πραγματικά μπορώ να το συστήσω σε όλους τους συναδέλφους θερμά να δραθούν τις ευκαιρίες με τέτοιες πρωτοβουλίες να δείχνονται αυτές οι ταινίες στις χώρες τους σε κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτό είναι μεγάλος πλούτος, μεγάλος εμπλουτισμός της πολιτιστικής ζωής. Μία επιθυμία θέλω να εκφράσω και το λέω κάθε φορά και θα την επαναλάβω και τώρα. Και ίσως Ντόρις μπορείς και εσύ αυτό να το διαβιβάσεις στα μέλη της ε, Ελλανοδίκου Επιτροπής. Ε, επί πολλά χρόνια βλέπουμε σοβαρές ταινίες με κάποιες εξαιρέσεις με πολύ σοβαρά και με βαθιές ρίζες προβλήματα και στο τέλος τέλος η έκβαση είναι πολλές φορές τραγική το τέλος της ταινία. Κάποιοι ενήλικες κιόλας έβγαζαν τα μαντήλια τους επειδή είχαν συγκινηθεί και είχαν με αυτόν τον τρόπο, πώς να το πω, ε, συμμετάσχει απόλυτα. Θα ευχόμουν όμως να είχαμε και μια κομμωδία. Κάποια έργα που θα ήταν κομμωδίες, που θα αντανακλούσαν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και που θα ήταν πιο εύθυμα, πιο χαρούμενα. Ξέρω ότι <clears throat> είναι η πιο δύσκολη τέχνη σίγουρα αυτή, αλλά πραγματικά θα εμπλούτιζε το κινηματογραφικό τοπίο στην Ευρώπη. Αν είχαμε και το έπαθλο Λουξ που θα απονεμόταν σε κάποιον κινηματογραφιστή που θα είχε γυρίσει μια τέτοια ταινία. Ας το πω έτσι μια κομμωδία. Μια εύθυμη κομμωδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γερκόνου. Τώρα θα πάρω λόγο και ήθελα να πω ότι Είχαμε και μια πολύ ωραία ταινία από την Ελλάδα, αλλά τελικά δεν κέρδισε. Κύριος Διακόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζήτω συγγνώμη πρώτα. Ίσως αυτό το θέμα θα παρατηρήσετε ότι είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό θα επικεντρωθώ. Η ταινία, οι ταινίες είναι η ζωή μου. Είμαι ηθοποιός και πάνω από 100 ταινίες γύρισα μέχρι σήμερα. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά αυτόν τον κλάδο, τον κινηματογραφικό και ξέρω και ποια είναι η δύναμη, η, η, η επιρροή και η δύναμη που μπορεί να ασκήσει μια ταινία και ο κινηματογράφος. Θαυμάζω λοιπόν μπορώ να πω εκείνους τους ανθρώπους που τους καίει η φλόγα, το πάθος για να συμμετάσχουν και να εκφραστούν. Και βλέπουμε όταν υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Τώρα για το ίδιο το θέμα που μας απασχολεί. Κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περίοδου ο κινηματογράφος στη Ρουμανία, ο πολιτισμός, τα πολιτιστικά θέματα, οι ταινίες είχαν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και επιρροή. Όλα αυτά υπό αυτό το κομμουνιστικό πλαίσιο. Είναι σαφές ότι έτσι το προσέγγιζαν και το κατανοούσαν οι πολίτες. Και όταν κάνουμε μια προβολή προοπτικά στη σημερινή κατάσταση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα δούμε ότι είναι ένας παράγοντας ε, κλειδί για τα όσα μπορούν και πρέπει να γίνονται και σε σχέση και με την ίδια την κρίση και τις ε, επιπτώσεις της ε, και τον σκεπτικισμό και την ε, ευρωσκεπτιστική τάση στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποστασιοποίηση ακριβώς όσον αφορά τις ταινίε. Αν μπορέσουμε με σοβαρό τρόπο να, να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες, αυτό θα ήταν σημαντικό για την Ευρώπη για παράδειγμα σε σχέση με την ταυτότητα και την ιστορία της κάθε χώρας, τις παραδόσεις της κάθε χώρας, να μπορούσαμε να συνδυάζαμε αυτά τα στοιχεία ώστε να γίνουν γνωστά στην Ευρώπη, να υπάρξει καλύτερη γνώση των πολιτών για τις άλλες χώρες και τους άλλους πολίτες και την ιστορία τους. Έτσι μπορούμε κάτι άλλο να μάθουμε και από πλευράς της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα. Με αυτό συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την κυρία Πακ και θα μπορούσα να συζητήσω τεχνικές λεπτομέρειες μαζί της πώς τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Όμως μια πρόταση μπορώ να κάνω ήδη τώρα. Το κλειδί για μια τέτοια πρωτοβουλία έγκυται πιστεύω στην κριτική επιτροπή. Εκείνοι έχουν την επιρροή και τις δυνατότητες στα χέρια τους. Θα έπρεπε λοιπόν να μεριμνήσουν οι κυριότεροι στόχοι να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τις ταινίε αυτές. Είναι λοιπόν σημαντικό σε κάθε φεστιβάλ, σε κάθε προβολή κινηματογραφικών ταινιών η Κριτική Επιτροπή είναι εκείνη που δίνει την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά σε αυτές τις ταινίες. Να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους πολίτες μέσα από αυτές ε, τις ε, πρωτοβουλίες. Η επιλογή θα πρέπει, η επιλογή θα πρέπει να γίνεται από τους Ευρωπαίους πολίτες λοιπόν ανεξάρτητα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την Doris για την μαχητική της παρουσίαση. Είναι πραγματικά έχει με μεγάλη επιτυχία η ιστορία του βραβείου Λούξ. Και είναι σημαντικό το ότι δόθηκε ε, η μάχη για αυτή την πρωτοβουλία. Δεν ήταν εύκολο, υπήρξαν επικρίσεις. Εν τω μεταξύ μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτό το, αυτές οι ταινίες και μέσα στο πλαίσιο του βραβείου Λούξ δίνει κάτι, δίνουν κάτι που δεν δίνουν άλλα μέσα όταν έχουμε υπόψη το τηλεοπτικό πρόγραμμα, πάντα υπάρχουν παράπονα ότι ήθιστε να μην παρουσιάζονται ευρωπαϊκέ ταινίε ε, στα τηλεοπτικά προγράμματα από τι άλλε χώρε. Με αυτό το βραβείο Λούξ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία την πολιτισμική ποικιλότητα και πολυμορφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να την παρουσιάσουμε και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι πραγματικά που να αξίζει τον κόπο. Και έτσι λοιπόν για μια ευρύτερη πρόσκληση σε σχέση με την ε, συμμετοχή σε αυτή την ε, πολυμορφία την ευρωπαϊκή θέλω να το ξανατονίσω αυτό ότι πρέπει να διαφημίσουμε αυτό το βραβείο Λουξ και να, το, να, να διαδοθεί η πρακτική αυτή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και έχουμε ένα στόχο να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ταινία. Να μην αφήσουμε τα ενία και τις πρωτοβουλίες στο Hollywood και το Bollywood. Είναι σημαντικό για τη διάχυση και διάδοση ευρωπαϊκών ταινιών λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτή, αυτό το βραβείο Λουξ να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χέλγα. Um, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να τοποθετηθώ για αυτό το θέμα. Ντόρες, δεν σε έχω γνωρίσει στο παρελθόν, γιατί με νεοκλεκτήσα, όμως χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ και ακούω τον ενθουσιασμό σου για τις ταινίε. Και ε, εγώ στο παρελθόν ε, έχω εργαστεί στον καλλιτεχνικό τομέα, σε μια καλλιτεχνική κοπερατίβα και συνεργαζόμασταν με νέους ανθρώπους και σε τοπικό επίπεδο ε, συνεργαζόμαστε με νέους και σε διεθνές επίπεδο συμμετείχαμε σε διάφορα προγράμματα και φεστιβάλ. Και σίγουρα αυτό στην πατρίδα μου, όχι μόνο στη δική μου περιφέρεια, αλλά και εθνικά. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε εδώ για τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων, αλλά θα έπρεπε να είμαστε πιο προδραστικοί για το πώς ε, χρησιμοποιούμε το βραβείο ε, παράλληλα με ανάληψη άλλων πρωτοβουλειών για τους νέους. Ε, δηλαδή, ε, ξέρω ότι εμείς έχουμε περιορισμένο χρόνο και πόρους, όμως ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι μια πρόκληση που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στην επιπροβολητισμού στο μέλλον, δηλαδή να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις δικές μας ικανότητες που συνεισφέρουμε εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γραμματικάκης. Και εγώ είμαι κινηματογραφόφιλος και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα ακούω για πρώτη φορά με τόσες λεπτομέρειες την ιστορία, την επιτυχία και το πάθος που συνοδεύει αυτό το βραβείο. Ε, θα κάνω λοιπόν ένα σχόλιο, αυτό είναι το σχόλιο, μια ερώτηση αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε και μία θα την έλεγα πρόταση. Το σχόλιο είναι, δεν ξέρω ακόμα, θα πω, τις, ε, τα κριτήρια της Επιτροπής της Ελλανοδίκου, αλλά ανησύσα λίγο, κυρία Πακ, επειδή μου είπατε ότι λίγο συγκλίνομαι με το Όσκαρ. Ελπίζω να μην είναι τελείως αλήθεια αυτό, γιατί εκεί θα βρει κανένας πάρα πολλές αδυναμίες. Αυτό που εμποδίζει τη διάδοση του βραβείου Λουξ και έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα στην Ευρώπη είναι ότι εμφανίζεται, ενώ μπορεί να είναι εξαίρετε οι ταινίε, ότι είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στους πολύπλοκους θεσμούς της, ότι είναι λίγο κατευθυνόμενη και αυτό αποθεί το μέσο θεατή. Επειδή προβληματίζομαι κι εγώ γι' αυτό, ε, εν καιρό ίσως σας γράψω, ίσως σα δω κάποιες ιδέες που έχω. Και στο τέλος ε, δεν τη λέω πρόταση. Έχετε σκεφτεί μήπως έπρεπε να επεκταθεί αυτό το σπουδαίο βραβείο, το πετυχημένο και σε άλλα φάσματα κινηματογραφικά, για παράδειγμα στο ντοκιμαντέρ που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για την ταυτότητα της Ευρώπης και ένα ιδιαίτερο είδος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Βέντα, τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ. Κυρία Πακ, ε, η παρουσίασή σας ήταν πραγματικά παθιασμένη και πιστεύω ότι το γραφείο Λουξ είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Αυτό μάλιστα υπογραμμίστηκε ήδη. δεν ε, μετράει μόνο ο νικητής, αλλά μετράει και η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Η πολυμορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού μας οδηγεί στο να χρειαζόμαστε τέτοια μέσα και εργαλεία για να προσεγγίζουμε τις ε, ταυτότητές μας. Σας ευχαριστώ κυρία Πάκ λοιπόν για αυτή την ε, παθιασμένη και ενθουσιώδη παρουσίαση και πρέπει να πω ότι συχνά στην Πολωνία έχουμε παρουσιάσει τις ταινίε που επιλέγονται για αυτό το φεστιβάλ και όταν παρουσιάσαμε αυτές τις ταινίε ήταν γεμάτες οι αίθουσε. δηλαδή υπήρχε το ενδιαφέρον από το κοινό και ελπίζω ότι έτσι θα συνεχίσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Σοντρόβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω κι εγώ με όλους όσους επένδυσαν την κυρία Πάκ Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη που η κυρία Πάκ θα συνεχίσει να ε, βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Ε, εγώ τον Δεκέμβριο θα είμαι στο screening για το ε, φεστιβάλ, για το Άιντα, στην Τσεχία. Αλλά τι γίνεται με την ε, ψηφοφορία ε, για τις ταινίες. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω και την άποψη των ε, θεατών, να ξέρουμε τι πιστεύουν και εκείνοι για τις ταινίε που παρακολουθούν. Αλλά κάποιες από τις προτάσεις που ακούστηκαν, για παράδειγμα για τα ντοκιμαντέρ, αν θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε και τις περιβαλλοντικές ταινίες ή τις παιδικές ταινίε. Υπάρχουν, υπάρχουν τέτοια φεστιβάλ κινηματογράφου στην Τσεχία και είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα που έχουμε από αυτά. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Πακ θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί το βραβείο Λουξ έχει αυτήν την μορφή, την ε, ε, ευρεία μορφή. Να επανέλθω στις παιδικές ταινίες είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ και είναι πολύ δύσκολο να ε, δημιουργηθούν ταινίε που είναι προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Κύριε Πάκ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχετε ενθουσιαστεί όλοι και με χαροποιεί αυτό, διότι χρειάζομαι τον δικό σας ε, ενθουσιασμό ε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε το βραβείο αυτό από το τμήμα επικοινωνίας. Ε, κάνατε κάποιες ερωτήσει. Να ξεκινήσω με την ε, Κριτική Επιτροπή. Η Κριτική Επιτροπή δεν μπορεί να αποτελείται από εμά. Η Επιτροπή επιλέγει ταινίε, που επιλέγει ταινίε και που μας τις προτείνει μας μπορούν να είναι άνθρωποι που ε, γνωρίζουν τις, ε, τις ταινίε της τελευταίας χρονιάς, που γι' αυτόν τον λόγο μπορούν και να τις προτείνουν και από, αυτές τις, από την τεράστια ποικιλία ταινιών επιλέγονται 10 ταινίε. Είναι όλοι ανεξάρτητοι. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι ανεξάρτητοι από όλες τις χώρες. Και από μας συμμετέχει πάντοτε ένας από αυτήν την ε, στην Επιτροπή αυτή. Δεν, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που, που είπε ο Έλληνα συνάδελφο, να συμμετέχουν περισσότερο οι, οι πολίτε. Το προσπαθούμε, αλλά η Κριτική Επιτροπή αυτή είναι η ειδική. Και σας δίνουν αυτές τις τρεις ταινίες και μετά εσείς είστε η μεγαλύτερη κριτική επιτροπή που έχει υπάρξει ποτέ για οποιοδήποτε κινηματογραφικό βραβείο και εσείς επιλέγετε ως εκπρόσωποι των πολιτών τον νικητή. Επειδή όμως είχαμε την ίδια αίσθηση με εσά ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι οι πολίτες, δημιουργήσαμε αυτά, αυτές, αυτή τη διοργάνωση Lux Film Days όπου όσοι προσέρχονται στις διοργανώσεις αυτές μπορούν να ψηφίσουν. Δεν γίνεται όμως να γίνεται αντίθετα. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την ε, αντίθετη πορεία γιατί οι πολίτες δεν ξέρουν τις ταινίε, γιατί αν τις ξέραν τις ταινίε δεν θα χρειαζόταν να υποστηρίζουμε εμείς τον υποτιτλισμό και τη διανομή. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία μόνο εφόσον οι πολίτες έχουν δει τις ταινίε αυτές. Και αυτό γίνεται με το Lux Film Days. Και στην περίπτωση της ταινία Band de Fille, της Γαλλίδας ε, σκηνοθέτηδας, ε, έγινε προβολή λοιπόν και την πρώτη μέρα μπορώ να σας πω ότι την παρακολούθησαν 25.000 άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία μπορείτε να το φανταστείτε 25.000 άνθρωποι είδαν αυτήν την ταινία και στις περισσότερες περιπτώσεις ε, υπήρχε ο υπότιτλος European Parliament is committed to culture Νομίζω ότι αυτό είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι η Κριτική Επιτροπή λοιπόν έχει τη, σύνθεση που θα έπρεπε. Το δεύτερο, κάντε μια, που, ακούστηκε, κάντε μια αστεία ταινία επιτέλους. Πάρα πολλοί άντρε μου έχουν πει και εμένα ε, κατά καιρού ότι μα κάθε φορά καθόμαστε και κλαίμε. Κάντε και κάτι να γελάσουμε λίγο. Καταλαβαίνω, αλλά ε, εγώ δεν είμαι στην κριτική επιτροπή. Ε, όταν το είπα κάποτε στην Κριτική Επιτροπή μου χαμογέλασαν ευγενικά αλλά μου είπαν «Ε, τι να κάνουμε. Είχαμε μια καταπληκτική ε, ελληνική ταινία, την Ακαδημία Πλάτωνος, μια χιουμοριστική ταινία με ένα εκπληκτικό, πολύ ενδιαφέρον θέμα, την αλβανική μειονότητα στην Ελλάδα. Ήταν πραγματικά καταπληκτική ταινία. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ήταν στις τρεις ταινίες στις τρεις ταινίε, αλλά τελικά δεν, δεν, δεν νίκησε. Ε, νίκησε τελικά η ταινία «Η Ξένη» ε, που αφορούσε τα εγκλήματα πάθους που νίκησε τελικά. Αλλά το διαφοροποίησαμε κι εμείς τη, τη διαδικασία μάλλον για αυτόν τον λόγο. Τώρα πλέον υποτιτλίζουμε και τις τρεις ταινίε. Αυτό δεν ίσχυε πέρσι. Ε, τα προηγούμενα χρόνια μάλλον. Ε, Υποτιτλίζαμε μόνο την ταινία που κέρδιζε το βραβείο. Τώρα, ποια κριτήρια ε, εφαρμόζονται. Μόνο ένα. Οι ταινίε αυτές θα πρέπει να έχουν προβληθεί σε κάποιο φεστιβάλ την προηγούμενη χρονιά. Ότι θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Δεν λέμε όμως ότι πρέπει να έχουν θέμα το άσυλο ή το τάδε θέμα. Αυτό δεν το κάνουμε και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε και να το κάνουμε. Οι ταινίε δεν γίνονται για, για, ακριβώς για, να μπορούν να προβληθούν στο κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα πολιτιστικό υπόβαθρο, υπάρχουν ε, κινηματογραφιστές. Αλλά ε, εξετάζουμε όλες τις ταινίε που έχουν κάποιο ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό που είπα για το Όσκαρ ήταν απλά μια παρατήρηση. Αυτό που είπα ήταν ότι η ταινία Ιντα που βρίσκεται στις τρεις δικές μας ταινίες για το Λουξ ε, έχει πάρει υποψηφιότητα για το Όσκαρ και είπα ότι ενδεχομένως υπάρχουν κοινά κριτήρια. Ε, και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε μια πολύ καλή κριτική επιτροπή που πραγματικά επιλέγει πολύ καλέ ταινίε. Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ ότι τα ντοκιμαντέρ πρέπει να τα συμπεριλάβουμε και ίσω θα έπρεπε να εξετάσουμε και τι παιδικέ ταινίε. Ισχύουν αυτά. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξή. Όταν δώσω κάτι. Όταν προσπαθήσω να. Ε, συγκροτήσω το διαγωνιστικό τμήμα ενό φεστιβάλ δεν, μπορώ να, δεν γίνεται να συμμετέχουν ταινίες ενηλίκων, παιδικές ταινίες, ντοκιμαντέρ ε, ταυτόχρονα. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ξεχωριστό βραβείο για όλα αυτά τα, για, για είδη ταινιών, αλλά ε, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα γι' αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε με την Κομισιόν στο μέλλον, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα τουλάχιστον δεν γίνεται να συμμετέχουν όλα αυτά τα είδη ταινιών γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη σύγκρισή τους. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προβολές σε σχολεία. Έχω πάει σε δύο γυμνάσια, Λύκια, όπου προβλήθηκαν οι ταινίες... Ε, η ταινία η Ξένη». Ε, σε ένα σχολείο λοιπόν ε, η, η ταινία αυτή αφορά τα εγκλήματα τιμής Και υπήρχε ένας καθηγητής ο οποίος πρόβαλε την ταινία αυτή μια, για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ε, και μάλιστα προσκάλεσε και ευρωβουλευτές. Ήταν πραγματικά φοβερό. Μπορώ να σας το πω και ως καθηγήτρια. Ήμουν κάποτε, πολύ παλιά. Είναι λοιπόν ένα παιδαγωγικό εργαλείο και διαπίστωσα ότι ακόμη και η Κομισιόν διοργανώνει τέτοιου είδους προβολές σε σχολεία ακριβώς για την, για την προβολή ε, των, ε, της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Λοιπόν, όλα αυτά που είπαμε εδώ ε, υπογραμμίζουν όλα αυτά που κάνουμε εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για, την, ε, για τα λουλούδια που μου δώσατε. Ε, και σας διαβεβαιώ ότι με πολύ μεγάλη χαρά θα εκτελέσω τα καθήκοντά μου αυτά, αλλά χρειάζομαι και τη δική σας υποστήριξη. Όπως ξαναείπα, στο DVD ή Video On Demand ή από 2 μέχρι 12 Δεκεμβρίου μπορείτε εδώ στον, στο, στο, στον κάτω όροφο να παρακολουθήσετε τις ταινίες αυτές και σας παρακαλώ ψηφίστε ψηφίστε κι εσείς για να έχουμε ψήφους από περισσότερο από το 1 τρίτο των ευρωβουλευτών που είχαμε μέχρι τώρα και νομίζω ότι στις 17 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια πολύ σύντομη μεν αλλά πολύ όμορφη εκδήλωση εορταστική 20 λεπτά ε, θα, θα διαρκέσει ε, πριν τις ψηφοφορίες το κάνουμε αυτό γιατί θα πρέπει, για να είναι γεμάτη αίθουσα τι να κάνουμε πρέπει να δίνουμε και κίνητρα σε ορισμένου συναδέλφου, αλλά εν πάση περιπτώσει να σα ξαναευχαριστήσω και βεβαίω όλα όσα ακούστηκαν εδώ και όλα όσα είπατε θα τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα στο μέλλον. Πριν να ευχαριστήσουμε και να αποχαιρετήσουμε την κυρία Πακ, θα ήθελα να δώσω στο συνάδελφο Γλέζο που ζήτησε το λόγο, αλλά δεν ξέρω για αυτό το σημείο θέλατε το λόγο. Παρακαλώ. Είχα καταλάβει ότι θέλατε το λόγο για κάτι άλλο συμφωνήσω απολύτως με την εισήγηση γύρω από τα θέματα που έθεσε και το περιεχόμενο και όλο το προβληματισμό που μας ε, είπε και που συμφωνώ απολύτως. Κάνω μία σημείωση, εδώ λυπούμε που αναφέρομαι στο πρόσωπό μου, αλλά ε, υπήρξα αντικείμενο ή θύμα αν θέλετε κινηματογραφικής μανίας. Ε, πριν από 70 χρόνια έγινε μια ταινία ε, για μένα, δεν ήθελα να προβληθεί, τελικά στη διάρκεια της Χούντας που δεν μπορούσα να πω γνώμη, την προβάλλανε παρά τη θέλησή μου. Και τώρα ακόμα δύο συνεργεία, ένα ελληνικό και ένα γαλλικό, με παρακολουθούν για να φτιάξουν ταινία για την, τον αγώνα που κάνω στο στο, στη σημερινή προσπάθεια για τη δημοκρατία. Ε, η πρότασή μου είναι όχι μια ταινία που θα πάρει το ροδίο Λουξ, αλλά προτείνω μια σούπερ Λουξ ταινία που θα έχει αντικείμενο τον Ευρωβουλευτή που αγωνίζεται μέσα από τη σκύλα και τη χάριδη του χρόνου να βρει τον τρόπο να εκφραστεί, να πει τη γνώμη του. Διότι με τα δευτερόλεπτα της γαλάζιας κάρτας, με τα δευτερόλεπτα του να μιλήσει και να γραφτεί. Και δεν θα μιλάς, μιλήσω για εισηγητές, μιλάω για τον Ευρωβουλευτή. Δεν έχει τη δυνατότητα να πει τη γνώμη του. Προβάλλουμε ταινίες πώς ένα πρόσωπο προσπαθεί να υπάρξει στη ζωή, πώς ένα πρόσωπο προσπαθεί να δείξει την ταυτότητά του. Ποιος θα φτιάξει, ε, υπάρχει ένα σκηνοθέτη εκεί, ένας, πώς θα φτιάξει τη ζωή, όχι, τον αγώνα του Ευρωβουλευτή να πει την άποψή του. Πώς, που δεν μπορεί, δεν τα καταφέρνει. Να και η απόδειξη η σημερινή. Εζήτησα να μιλήσω πριν από την ημερήσια διάταξη. Μου απαγορεύτηκε. Πρωτοφανέ. Ζητάει ένα ευρωβουλευτή να μιλήσει πριν από την ημερήσια διάταξη και του απαγορεύεται να μιλήσει. Αρχίζει η ομιλία. Σηκώνω κάρτα, δεν μου δίνεται ο λόγο. Δεν μπορώ να την καταλάβω εντελώ αυτή την άποψη και αυτή την αντίληψη. Τελικά, σας καταγγέλω ότι έχετε καρφώσει στον κάφκασο της εξουσίας τη δημοκρατία. Και μην ξεχνάτε ότι η βοηθή του Ερμή για το κάρφωμα του Προμηθέα και το κάρφωμα της δημοκρατίας τώρα ήταν η βία και το κράτος. Λοιπόν, σας πληροφορώ και αγωνίζομαι, δεν πρόκειται να σας αφήσω ίσως. Όσο ζω και όσο υπάρχω θα ακούτε τη φωνή μου δεν θα πρόκειται να τη δεσμεύσετε μέσα στα χρονικά όρια στραγγαλισμού των δευτερολέπτων και των μισών λεπτών. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, λυπάμαι που εσείς αξιολογήσατε με αυτόν τον τρόπο τη στάση της Προεδρίας που δεν ήταν καθόλου αντιδημοκρατική. Όταν μου είπατε ότι θέλετε να μιλήσετε είχαμε ήδη ξεκινήσει τη συνεδρίαση ζήτησα να μάθω για ποιο θέμα και δεν μου εξηγήσατε. Δεν ε, ήξερα εγώ για ποιο θέμα θέλετε να μιλήσετε. Είχαμε ήδη εδώ τη συνάδελφο Ντόρις Πακ, ε, ήταν για αυτό το θέμα. Εγώ νόμιζα ότι θέλατε να πάρετε το λόγο ε, στη συνέχεια. Αν σας παρερμήνευσα, με συγχωρείτε, όμως σας μην εκτοξεύουμε εδώ διάφορες κατηγορίες περί αντιδημοκρατικού, δικτατορικού κτλ. Ξέρω ότι δεν ε, υπάρχει εδώ τέτοια βούληση καταναγκασμού. Πάντως προσωπικά σας ζητώ συγγνώμη αν δεν σας κατάλαβα καλά. Δεν ήταν πολύ σαφής ο τρόπος με τον οποίο ζητήθηκε ο λόγος. Πάντως σέβομαι το θέμα που θέτετε Πάντως, ε, ειλικρινά αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται με την κυρία Πάκος ε, συντονίστρια. Για το βραβείο Λούξ, εσείς θέτετε ένα θέμα ενδιαφέρον. Ε, εδώ συζητάμε το θέμα της δημοκρατίας και μέσω της κινηματογραφικής γλώσσας. Εμείς θέλουμε να... Τώρα εδώ, αν μας είπατε ότι πρέπει να οργανωθούμε για να γνωστοποιήσουμε το τι συμβαίνει εδώ, δεν ε, ξέρω αν αυτό μπορούμε να το προτείνουμε επίσημα για να υπάρχει ένα βραβείο του Κοινοβουλίου. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον για τους πολίτες ε, να μάθουν πώς εμείς δραστηριοποιούμαστε εδώ. Αν κάποιος σκηνοθέτης θέλει να τον αναλάβει μπορεί να ήταν μια καλή ιδέα. Όμως ε, αυτά που μας είπατε δεν αφορούν το βραβείο Λουξ το βραβείο Λούξ δεν μιλά για μας, μιλά για διαφορετικά θέματα, για την ε, δημιουργία, για ευαίσθητα θέματα που αφορούν τους Ευρωπαίους. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό το θέμα μπορεί να τεθεί στην Επιτροπή Πολιτισμού. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ την Doris Σπάκ, για αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει και για το πώς σκοπεύει να το διαδραματίσει. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα Μαρσελέο Ρωσέτη Κίτρικ για το έργο τους, για τη δουλειά τους ε, και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και μαζί σου και μαζί μας. Τρίτον, νομίζω ότι μπορούμε να προωθήσουμε ε, και εμείς το βραβείο Λουξ, τη γνώση για το βραβείο Λουξ και επίσης να γνωστοποιήσουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στις ενώσεις ε, των παραγωγών και των διανομέων. Δηλαδή και στη χώρα μου υπάρχει μια τέτοια έλλειψη γνώσης. Εδώ συμφωνώ με τη συνάδελφο Πέτρα ε, για την αξία που έχουν ε, οι μικροί κινηματογράφοι ε, γνωστοποιούν τις ταινίες άλλων χωρών και στη Ρώμη Υπάρχουν ε, πολλοί μικροί κινηματογράφοι που θέλησαν ε, να διαδώσουν και να παρουσιάσουν αυτές τις ταινίε. Και νομίζω ότι για το θέμα της Κριτικής Επιτροπής σίγουρα θα υπάρχει ε, μια περιτροπή των μελών. Θα ήταν καλό αυτό για να υπάρχει και διαφάνεια. Όμως εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα γιατί υπάρχει εδώ μια ένδειξη, δηλαδή να συζητάμε για θέματα που είναι ευαίσθητα αλλά θέλουμε να υπάρχει αυτονομία και ανεξαρτησία της Κρητικής Επιτροπής. Εσείς ε, ξέρετε ότι στις 17 Δεκεμβρίου θα είναι η ολοκλήρωση της προετοιμασίας μας, γιατί κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας επίσημα πριν από την ψηφοφορία, ε, όπου θα περιβρισκόμαστε όλοι, θα ε, προσκληθούν οι τρεις φιναλίστ και τότε θα ανακοινωθεί και ο νικητής και συνήθως ε, οι νέοι σκηνοθέτες παίρνουν το λόγο στην Ολομέλεια και πάντοτε είναι πολύ συγκινημένοι. Εγώ θυμάμαι και τον Αντέα Σέγκετς όταν παρουσίασε την ταινία του. Έτσι λοιπόν ε, θα υπάρχουν συμμετοχές και καλού όλους τους συναδέλφους ε, να έρθουν σε επικοινωνία με τους συναδέλφους τους από τις άλλες επιτροπές γιατί θέλουμε αυτό το βραβείο να είναι ένα βραβείο του Κοινοβουλίου, όχι της δικής μας επιτροπής μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Πάκ και καλή επιτυχία. Allora, grazie Doris. Noi penso che adesso dobbiamo... Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με την ημερησία διάταξη. Θα περάσουμε τώρα στην έκθεση που έχει αναλάβει ο συνάδελφος Βέντα για το Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ουσιαστικά για την έκθεση πρωτοβουλία. Ξέρετε ότι πρόκειται για μια σημαντική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάιο για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο και την ε, ανάπτυξή του. Επίσης αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας αυτό στην ψηφιακή εποχή. Πρόκειται για μας για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα μας πει ο εισηγητής ποιες γραμμές θέλει να ακολουθήσει και κατόπιν θα έχουμε συζήτηση με τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα θέμα, μπορώ να πω, που κατά την έναρξη της συνεδρίασης για το βραβείο Lux ε, έχω την τιμή συνάδελφοι να είμαι εισηγητής για το θέμα αυτής της έκθεσης για την ε, κινηματογραφική βιομηχανία και σε σχέση με μια ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά. Είναι ένα από τα θέματα κλειδιά για την δική, δική μας ε, Επιτροπή. Οι ταινίε είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την διάχυση της πολιτισμικής πολυμορφίας. Να μάθουμε κάτι και για τους ε, γείτονές μας. Κατά την τελευταία περίοδο είχαμε μία έκθεση για αυτό το θέμα η μετάβαση δηλαδή από τις ε, κανονικές ε, ταινίες στις ψηφιακές, ε, στην ψηφιακή εποχή. Η πρόταση λύσεων που θα επέτρεπε στους θεατές να έχουν την βέλτιστη πρόσβαση σε σχέση με αυτά τα πολιτισμικά προϊόντα και όσον αφορά την διάχυση και την προώθηση ταινιών, ευρωπαϊκών ταινιών. Οι ευρωπαϊκές ταινίες σε σχέση με το ποσοστό τους είναι μόνο ένα τρίτο των εισιτηρίων σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες και είναι στον αριθμό περίπου των 1.000 ή 1.300. Οι περισσότερες ταινίες ε, προβάλλονται στις χώρες τους και σπάνια προβάλλονται σε άλλες χώρες. Σε σχέση με τις ΗΠΑ, 800 ταινίες ετήσια παράγονται. Όμως η ε, ε, διάχυση, η διάδοση, η προαγωγή αυτών των ταινιών είναι πολύ πιο επιθετική και παραγωγική σε σχέση με τον τρόπο που ε, λειτουργεί η Ευρώπη. Πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά μας λοιπόν. Αυτό αποτελεί και ένα μέρος της δημιουργίας της ευρύτερης της μίζωνος Ευρώπης. Είναι απόδειξη ότι κάτι παραπάνω πρέπει να κάνουμε για να αυξηθεί ο αριθμός εκείνος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ταινίε. Μέσα στο πλαίσιο, για παράδειγμα, της διασυνοριακής συνεργασίας, να προβάλλονται περισσότερες ευρωπαϊκές ε, ταινίε. Και είναι και ένα θέμα χρονικής ε, συγκυρίας που θα βρίσκονται αυτές οι ταινίε ε, στην πρώτη γραμμή. Κάποιες μελέτες όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν ότι 70% στο διαδίκτυο παρακολουθούν τέτοιες ταινίες, κατεβάζοντάς τις είτε παράνομα είτε νόμιμα. Και κατά 40% χρήστες των ε, smartphones και των ε, ταμπλετών και υπολογιστών με τον ίδιο τρόπο ε, δρούν. Ίσως αυτό φαίνεται κάτι το προσδοκητό όμως υπάρχει το ενδιαφέρον για τα κινηματογραφικά προϊόντα και η επιλογή των ταινιών πολλές φορές είναι πιο περιορισμένη και όλα αυτά δείχνουν ότι ο κινηματογραφικός τομέας μπορεί να αυξήσει τα έσοδα του χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες του διαδικτύου σε σχέση με την διαθεσιμότητα και την προβολή των ταινιών αυτών, των προϊόντων αυτών των τηλεοπτικών, ώστε να φτάνουν σε μεγαλύτερο αριθμό θεατών και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ε, οι α, πόροι ώστε να υπάρξει αντίστοιχη διαφήμιση. Ακόμα όμως και αν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τέτοιες ταινίε νόμιμα μέσα στα α, νόμιμα πλαίσια. Αν κάποιος ε, θέλει να δει μια τέτοια ταινία πρέπει να αναμείνει, να περιμένει μήνες και μήνες ε, μέχρι ότου να μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια τέτοια ταινία. Και αναφέροντας το αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η τηλεόραση είναι το μέσο εκείνο που χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και η πλειοψηφία σε σχέση με τις ταινίε που προβλήθηκαν, που ήταν σε σχέση με την ευρωπαϊκή τους προέλευση, ε, ένα ποσοστό ήταν εθνικές ε, ταινίε, ένα άλλο από άλλες ευρωπαϊκές ε, χώρες. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το σύνθετο χαρακτήρα και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει και η δυνατότητα του βίντεο μετά από αίτημα ε, πρέπει να αυξηθεί και η ελαστικότητα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των ταινιών δηλαδή για το πότε και πόσα θα διατίθεται μια ταινία σε τέτοιου είδους προβολές και όταν βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο χρησιμοποιείται για τις κινέζικες ταινίες και τις ταινίες των ΗΠΑ, ο ανταγωνισμός ήδη έχει αυξηθεί και αυξάνεται. Το πρόβλημα είναι της χρηματοδότησης, είναι χρηματοδοτικό. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, όπως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, για τον Κινηματογράφο, ώστε 1,2 δις να μπορεί να, να διατίθεται αιτήσια. και βλέπουμε ότι από πλευράς της, ε, του προγράμματος Creative Europe δημιουργική Ευρώπη, θα πρέπει να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στον αυξανόμενο αριθμό θεατών που ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές αυτές ταινίες ως προϊόντα. Να υπάρχει δυνατότητα αύξησης και διάχυσης των προϊόντων αυτών. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στοχεύει στην παραγωγή των ταινιών αυτών και όχι για την αύξηση των ενδυνάμει θεατών τελικά που θα ήταν οι αποδέκτες αυτών των προϊόντων. Και πρέπει να δούμε ότι αυτός είναι ένας ρόλος κλειδί που έχει πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον. Διότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτές τις 800 σε ένα διάστημα 7 ετών η πλειοψηφία αυτών των κονδυλίων θα υποστηρίζει την υποστήριξη διάδοσης των ευρωπαϊκών αυτών ταινιών εκτός της χώρας παραγωγής τους η δημιουργία αυτού του φόρουμ λοιπόν, αυτού του βήματος ως χώρου είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, για το πώς ε, εθνικά χαρακτηριστικά, ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά μπορούν να είναι αλληλοσυμπληρούμενα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αναζωογόνηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας, διότι πολλοί κινηματογραφιστές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για να εξεύρουν κονδύλια. Και ο υποτιτλισμός, οι μεταφράσεις θα είναι ένας τρόπος για να είναι πιο προσπελάσιμες αυτές οι ταινίες. Ο υποτιτλισμός είναι ένας τρόπος να είναι πιο κατανοητές, να γίνονται πιο εύληπτες και κατανοητές αυτές οι ταινίες σε μια γλώσσα που ε, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είναι κατανοητή. Και αυτό έχει επιπτώσεις και σε σχέση με την ε, αντίληψη και που μπορεί να προαχθεί από πλευρά θεατών για το ποιο είναι το μήνυμα μια ταινία. Ο υποτιτλισμός λοιπόν είναι πολύ φθηνότερο σύστημα από ότι κατά την προηγούμενη περίοδο που δεν υπήρχαν ψηφοποιημένα, ψηφιοποιημένα προϊόντα και είναι δυνατόν έτσι να δραστηριοποιηθούμε πιο παραγωγικά. Και είχα και συμμετάσχει σε ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα για τον υποτιτλισμό που η νόμιμη, η νόμιμη δυνατότητα υποτιτλισμού θα ε, την χάνει ευρύτερη διάδοση. Αυτό θα δημιουργήσει και σε λιγότερο δαπανηρές ε, διαδικασίε ε, σε φθηνότερα προϊόντα. Ο υποτιτλισμός online στο διαδίκτυο είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι απόλυτα νόμιμο και έτσι πρέπει λοιπόν να υπάρξει η ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας. Ένα άλλο στοιχείο στην έκθεσή μου που θα έχει σημαντική ιδιαίτερη σπουδαιότητα θα είναι η εκπαίδευση για τις ταινίες και τα μέσα που θα ξεκινά από τα πρώτα χρόνια η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η παιδεία ευρύτερα δίνει την δυνατότητα να μπορούν με κριτικό πνεύμα να αξιολογούν και να παρακολουθούν ε, οι πολίτες ε, αυτά τα προϊόντα. Και εκπαιδεύοντας τους νέους με κριτικό πνεύμα να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, αυξάνοντας τις γνώσεις, τους, αυξάνει και την δυνατότητα να γίνονται υπεύθυνοι καλοί πολίτες στη Γαλλία, στη Δανία για παράδειγμα, που είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα η εκπαίδευση για τα μέσα, δείχνει αποδεικνύει ότι οι νέοι θεατές που συμμετείχαν σε τέτοιου είδους προγράμματα συνειδητά προτιμούν τις ευρωπαϊκές ταινίες όσον αφορά τον ρόλο των κινηματογραφικών προβολών των φεστιβάλ και του βραβείου Λούξ έχουν κύριο ρόλο να διαδραματίσουν εκπαιδεύοντας τους νέους Ευρωπαίους πολίτες σε σχέση με αυτή την πολιτισμική συνιστόσα και επίσης μπορούν να στο Κάρλο Βιβάρι στη Βενετία, στο Βερολίνο, στις Κάνες τα πλαίσια αυτών των φεστιβάλ για την επιλογή και την βράβευση ταινιών που έχοντας αποκτήσει αυτό το κύρος οι ταινίε αυτές διευκολύνονται μετά στην προβολή και στην ε, διάδοσή τους συνοψίζοντας θα ήθελα να αναφέρω τα εξή. οι νεαροί θεατές ε, βρίσκονται σε υπεύθυνη θέση αποφασίζουν εκείνοι υπεύθυνα τι θέλουν να δουν επιλέγουν είναι σημαντικό όμως ε, να μπορούν μέσα από τις δυνατότητες που τους προσφέρονται να δράσουν είναι με κριτικό πνεύμα ε, ε, δρούν σε πολύ κρίσιμες περιστάσεις ε, η παραγωγή για τη δημιουργία αυτών των ταινιών. Όμως η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια έχει το δυναμικό να προσελκύσει εκατομμύρια θεατών. Η άθικτη, για παράδειγμα, ως ταινία, που ήταν η, πιο δημοφιλής ταινία και 20 εκατομμύρια θεατές την παρακολούθησαν κατά το πρώτο διάστημα μετά την διανομή της. Ήταν κάτι αξιοθαύμαστο. Ήταν η πιο κερδοφόρα ταινία εκτός, ε, ε, από, εκτός των αμερικανικών ταινιών που προβάλλονται στα αγγλικά και έτσι έτυχε της προσοχής εκατομμυρίων θεατών παγκόσμια. Είναι κάτι το σημαντικό αυτό. Βλέπουμε εδώ ε, τις ε, διαχωριστικές γραμμές ε, που καθορίζουν τις δυνατότητες. έχω προθυμότητα, προθυμία να συνεργαστώ και να ακούσω τις απόψεις σας, ώστε να υπάρξει συνεργασία όπως πρέπει με τους σκιώδεις εισηγητές. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν για αυτή την προσπάθεια και την Επιτροπή των Περιφερειών που συμμετέχει και είναι παρούσα και για την ε, αναφορά για το βραβείο Λούξ. Θα πρέπει σε workshops, σε σεμινάρια να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στις 18 Νοεμβρίου στις 12 ε, θα υπάρξει αυτή η πρόσκληση. Θα έχουμε ε, προσώπους από την, τον, την Ένωση Κινηματογραφιστών και άλλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε, επειδή υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά σημεία που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν και έχουν υπογραμμιστεί και από εσά και φυσικά είναι χρήσιμα για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση της εκθεσής σας. Θα ξεκινήσει και μια συζήτηση με τους συναδέλφους. Φυσικά γνωρίζω ότι και εμείς ε, επιθυμούμε η ιδιαιτερότητα του κινηματογράφου να διατηρηθεί και να υπάρχει πάντοτε σεβασμός του πολιτισμού και της κινηματογραφικής κληρονομιάς που θα πρέπει να υπάρχει ακόμη και στα σχολικά προγράμματα. Αυτή είναι μια εισαγωγή και κατόπιν θα υπάρχουν ε, και ε, ακόλουθα θέματα όπως θα είναι η ενίσχυση της διανομής, ε, διάβριση του κοινού αλλά και οι απαραίτητες ικανότητες και η αλυσίδα ταξιας Καταρχήν να δώσουμε το λόγο στην Πέτρα που τον έχει ζητήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Βέντα για την παρουσίασή του. Η πρόθεση των ταινιών, το συζητήσαμε και για το βραβείο Λουξ, ε, ένας από τους σημαντικούς τομείς της πολιτικής μας πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, υπάρχουν δύο πλευρές ε, του ίδιου νομίσματος που αναδεικνύονται. Αφενός δηλαδή πρόκειται για μια προώθηση οικονομική ηθικού χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά βεβαίως η πρόθεση των ταινιών έχει και έναν δημιουργικό χαρακτήρα και έναν υψηλό πολιτισ... μια υψηλή πολιτιστική αξία. Οπότε γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι είναι σημαντικός ο τομέα. Χρήματα και κονδύλια για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την παραγωγή αλλά όχι για την εμπορία των ταινιών αυτών, για το marketing και στις ΗΠΑ για παράδειγμα τα χρήματα που ξοδεύονται μόνο για το marketing ε, είναι το 1 τρίτο ενώ στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι 10%. Και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το τομέα, πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, ώστε οι ταινίε που γυρίζονται να φτάνουν και στο κοινό στο, οποίο ε, απευθύνονται. Θεωρώ επίσης ότι κάθε αξιοποίηση ε, ταινιών ε, όπου κανείς μπορεί να αποκομίσει και εισόδημα θα πρέπει να διέπεται και από ένα σύστημα ε, συμμετοχής και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ε, προσαρμοστεί και στην ψηφιακή εποχή. Στη Γερμανία προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο και αυτή τη στιγμή έχουμε μια ε, δικαστική διαμάχη σε εξέλιξη και το κέντρο, το θέμα της ήταν ε, ε, η άποψή μου είναι ότι αυτό, όσοι, εν πάση περιπτώσει, βγάζουν χρήματα από τη διανομή των ταινιών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα ότι οι άνθρωποι που παράγουν τις ταινίες θα μπορούν να συνεχίσουν να φτιάχνουν και άλλες ταινίες. Έχουμε και ένα άλλο, προβλήμα, ένα άλλο πρόβλημα, στη Γερμανία τουλάχιστον ήταν πολύ έντονο αυτό. Δύο προσπάθειες είχαμε στο παρελθόν. Η κινηματογραφική κληρονομιά, ε, αυτά που είχαν ε, δημιουργηθεί για την, για την τηλεόραση να γίνουν δημόσια προσβάσιμα. Είχαν προσπαθήσει δύο τηλεοπτικά κανάλια να φτιάξουν μία ε, βιβλιοθήκη, ε, ψηφιακή βιβλιοθήκη και, τα, και οι δύο προσπάθειες είχαν απαγορευτεί από την Επιτροπή Καρτέλ και τώρα έχουμε ξαφνικά το Netflix μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία δηλαδή η οποία προσφέρει το δικό της περιεχόμενο χωρίς καμία επιτροπή για την καταπολέμηση των καρτέλ να μπορεί να τη σταματήσει. Οπότε νομίζω ότι ε, και σε αυτό το τομέα ίσως θα έπρεπε να, ε, να εξασφαλίσουμε ότι δεν εμποδίζουμε την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα και ότι δεν αφήνουμε απλά το όλο ζήτημα αυτό στους Αμερικανικούς Ψηφιοποίηση κινηματογραφικής κληρονομιάς είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και γνωρίζουμε όλοι ότι στα αρχεία όχι μόνο των τηλεοπτικών καναλιών αλλά και των κινηματογραφικών αιθουσών υπάρχουν θησαυροί που όμως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν για πάντα αν δεν ψηφιοποιηθούν άμεσα. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για αυτό το έργο και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πολύ γρήγορα λύσεις και υποστήριξη και χρηματοδοτική υποστήριξη γιατί αλλιώς οι ταινίες αυτές θα χαθούν για πάντα και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ κρίμα να επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, όσον αφορά, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη διαφορετική συμπεριφορά των καταναλωτών. Φυσικά είναι πάρα πολύ ωραίο να παράγει κανείς μια ταινία και, να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι να τη βλέπουν στην, αίθουσα. Ξέρουμε όμως ότι... Ε, αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Γιατί ξέρουμε ότι μετά το λανσάρισμα μια ταινία στην κινηματογραφική αίθουσα, μετά από πολύ λίγο χρονικό διάστημα, υπάρχει ανάγκη η ταινία αυτή να βγει και σε DVD ή σε video on demand. Αν δεν αλλάξουμε την στάση μα, θα πρέπει να δούμε, θα πρέπει βεβαίω να δούμε ε, ε, τι επιπτώσεις θα, θα υπάρξουν για τις κινηματογραφικές αίθουσες αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις τάσεις που υπάρχουν στην αλυσίδα αξία, της εξελίξης που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και να λάβουμε υπόψη μας όλες τις επιπτώσεις που ενδεχομένως βεβαίως θα προκύψουν για τις κινηματογραφικές αίθουσες αλλά και για τους ε, παραγωγούς και για τους, ε, ε, καλλιτέχνε. Θυμάμαι μια πολύ ωραία εκδήλωση που είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο όπου ο μεγάλος Βιμ Wenders μας είχε εξηγήσει ότι το να παρακολουθεί κανείς ταινίες είναι κάτι που πρέπει να μάθει κανείς. Γιατί οι άνθρωποι ε, και τα παιδιά από το σχολείο πρέπει να μάθουν, να διαβάζουν, όχι μόνο να παρακολουθούν, να βλέπουν μια ταινία, αλλά να τη διαβάζουν κιόλας. Οπότε θεωρώ κι εγώ ότι πρέπει να είναι σημαντικό στοιχείο της ε, εκπαίδευσης, της σχολικής εκπαίδευσης, των σχολικών προγραμμάτων, γιατί συνδέεται και με τη σημασία του πολιτισμού και οι κινηματογράφοι μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό σημείο εξωσχολικής εκπαίδευσης όπου μπορεί να υπάρξει πολύ καλή συνεργασία με τα σχολεία και ίσως είναι και ένας τρόπος αυτός να ξαναενισχύσουμε τους κινηματογράφους ώστε να ξαναπάνε και οι νέοι άνθρωποι στον κινηματογράφο. Τώρα, ε, φυσικά σημαντικό είναι ε, ότι και συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να προωθηθεί ποιότητα και η του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Νομίζω ότι οι προτάσει της Κομισιόν είναι πάρα πολύ καλέ, Θα τι επεξεργαστούμε και νομίζω ότι θα τι βελτιώσουμε και λίγο παραπέρα. Χαίρομαι που θα έχουμε μια πολύ καλή ε, συνεργασία με τον εισηγητή και με τους χειώδεις εισηγητές και νομίζω, είμαι σίγουρη δηλαδή, ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να συντάξουμε μια έκθεση η οποία θα εξυπηρετεί ακριβώς την προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στην Ευρώπη. Και σας παρακαλώ να μην με παρεξηγήσετε ε, αν σηκωθώ τώρα, αν με δείτε να σηκώνομαι και να φεύγω. Δυστυχώς πρέπει να πάω σε μια άλλη ε, εκδήλωση, αλλά θα έχουμε σίγουρα και στο μέλλον ε, και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε το θέμα αυτό περισσότερο. Ευχαριστώ. Πέτρο Και τώρα η Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο εισηγητή. Θέλω μόνο σύντομα να αναφέρω το εξή. Είναι απόλυτα σωστό ότι πολύ λίγα χρήματα δίνουμε για την διαφήμιση αν συγκρίνουμε με το Hollywood. Κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Φυσικά συμμερίζομαι και τον στόχο ώστε να υπάρξει καλύτερη προσπελασιμότητα και καλύτερη διάχυση των ευρωπαϊκών ταινιών, ε, πιο εύκολη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές ταινίες και ευρύτερη πρόσβαση και στο διαδίκτυο. Αλλά πρέπει και αδειμονώ να δούμε, να, να δούμε τις προτάσεις. Πρέπει να απαντήσουμε το ερώτημα όταν θα υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση διασυνοριακά, πράγμα που επιθυμούμε, πώς θα χρηματοδοτούνται οι ευρωπαϊκές ταινίε μελλοντικά, διότι συνδέονται σήμερα με την εδαφικότητα, με το θέμα της χρηματοδότησης των παραγωγών. Όταν διασυνοριακά θα προσφέρονται τέτοιες υπηρεσίες, δεν θα ταιριάζει αυτό το πρότυπο πια. Πρέπει να προβληματιστούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Διασυνοριακές άδειες που θα χορηγούνται ευρωπαϊκές άδειες που θα εκδίδονται. Το ερώτημα είναι τι θα κοστίζουν, τι θα στοιχίζουν όλα αυτά για αρκετές χώρες ε, σε σύνδεση, τι θα στοιχίζουν αυτά. Ή αν μπορεί να υπάρχουν ειδικέ άδειες ε, για το ε, διαδίκτυο, για βίντεο και πρέπει να δούμε αυτές τις, αυτά τα θέματα πιο εξειδικευμένα. Μέσα από αυτό το πρόβλημα είναι το ερώτημα, προ, προβάλλει το ερώτημα πώς θα χρηματοδοτούνται οι ευρωπαϊκές ταινίες. Με τη δημόσια χρηματοδότηση αυτό από μόνο του δεν επαρκεί. Πρέπει να ευρεθεί το σωστότερο πλαίσιο χρηματοδότησης και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον συνάδελφο Βέντα και να του πω ότι τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή του. Εγώ όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό πάντα βλέπω κάποιες ταινίε που θα ήθελα να παρακολουθήσω και όταν φτάνω στη χώρα μου, στην Ισπανία, τελικά να αδύνατο να τις δω γιατί δεν διανέμονται. Επομένως μου φαίνεται πολύ σημαντική αυτή η ιδέα να ε, επιμείνουμε στο θέμα της διανομής. Νομίζω ότι για μένα είναι πιο σημαντικό το θέμα της διανομής από της παραγωγής. Πολλές φορές έχουμε μεγάλη χρηματοδότηση για παραγωγή ταινιών που κατόπιν κανένας δεν βλέπει και δεν είναι ενδιαφέρουσες, ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες ταινίες πολύ ενδιαφέρουσες που δεν μπορούν ε, να τις δούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει κυρίως να δώσουμε έμφαση στη διανομή. Ο συνάδελφος Βέντα μίλησε και για τον αποτεκλισμό. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα ιδιαίτερα η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει με φτηνό τρόπο να μπορούμε να αποτεκλήσουμε τις ταινίε σε πολλές γλώσσες. Εγώ είμαι εντελώς αντίθετος στις ποσοστώσεις ανάλογα με τις γλώσσες. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει στην Καταλωνία όπου η κυβέρνηση επιβάλλει κάποιες ποσοστώσεις, ε, δηλαδή για να υπάρχουν συγκεκριμένες ταινίε στα καταλλανικά. Και αυτό έχει απορριφθεί από την Κομισιόν, αλλά συνεχίζει η κυβέρνηση τη Καταλωνία να επιμένει. Έχουμε μια πρόκληση ενωπιών μα, είναι αλήθεια. Και κάθε φορά δυστυχώ οι άνθρωποι πηγαίνουν όλο ένα και λιγότερο στον κινηματογράφο και περισσότερο αγοράζουν DVD, και όμως βλέπουμε ότι σήμερα περιορίζεται και το DVD και περισσότερο επιλέγουν το διαδίκτυο για το θέμα της πειρατείας, των παράνομων αντιγράφων, το να κατεβάζει κανείς δωρεάν ταινίες, όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε. Νομίζω ότι πολλοί νέοι που δεν θα μπορούσαν να κλέψουν ένα πορτοκάλι από το σούπερ μάρκετ, βλέπουν αντίθετα πάρα πολύ φυσιολογικό να κατεβάσουν παράνομα μία ταινία από το διαδίκτυο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία εκστρατεία για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την πειρατεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Σολβένη. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε πρώτη φορά εκλεκτικά εδώ στο Κοινοβούλιο. Ίσως ε, θα ήταν καλύτερο λοιπόν να μου δίνετε το λόγο αφού έχουν μιλήσει άλλοι πιο πεπειραμένοι συνάδελφοι. Όμως έχω εργαστεί για έναν τηλεοπτικό σταθμό για έτη που ήταν και εξειδικευμένο στην παρουσίαση ευρωπαϊκών ταινιών και επομένως μπορώ να καταλάβω τη σημασία του θέματος αυτού. Σας ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία αυτή. Όταν ήμουν νέος ε, πάντοτε ήθελα να με καταλαβαίνουν και τώρα που δεν είμαι και τόσο νέος εξακολουθώ να επιθυμώ το ίδιο και θα ήθελα να περάσω αυτό το μήνυμα και στα δικά μου παιδιά. Επομένως, ε, για να είμαι πιο κατανοητός, θα επικεντρωθώ σε ένα ζήτημα που αφορά το επιγραμμικό περιεχόμενο. Πάντοτε θα είναι άνθρωποι που πηγαίνουν στον κινηματογράφο γιατί τους αρέσει ο κινηματογράφος. Όμως, Χωρίς ε, το διαδίκτυο δεν μπορούμε να περάσουμε στις νεότερες γενιές αυτή την ε, πτυχή πολιτισμού. Η ομιλία του κυρίου Βέντα Άκουσα μάλλον τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις ε, και ε, μου φάνηκε σαν να έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κινηματογράφο, όμω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αλλά ε, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Εγώ μπορώ να δω αυτή την αντίφαση και θα ήθελα να το παρουσιάσω αυτό ως πρόκληση. Δεν έχω εντοπίσει αυτό το πρόβλημα στην έκθεση, αλλά θέλω να αναφερθώ σε αυτό ω πρόκληση. Οι Ευρωπαϊκέ ταινίε ποτέ δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικέ με τι αμερικανικέ ταινίε. Από μια εντελώ επιχειρηματική σκοπιά, ούτε καν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και να μπούμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί αν το προσπαθήσουμε θα χάσουμε πολλά χρήματα. Και αυτό είναι μια παρεξήγηση που υπάρχει. Ίσως αυτό που θα έπρεπε να περάσουμε ως μήνυμα είναι αυτή η ευαισθησία στις σχολές μας. Πρέπει να προβαλούμε περισσότερο τις ευρωπαϊκές ταινίε, να τις προβάλλουμε περισσότερο στα σχολεία μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ζήτηση για τις ευρωπαϊκές ταινίε και Το αν παρακολουθούμε αυτές τις ταινίε ε, στους κινηματογράφους ή online, στο διαδίκτυο, είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Η Γερμανία βρίσκεται σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Έχει μια τεράστια εγχώρια αγορά με 100 εκατομμύρια ενδυνάμοι θεατές ενώ τα περισσότερα άλλα, άλλα κρατημέλη είναι μικρότερες αγορές. Και θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο πώς θα έχουμε περισσότερο διαθέσιμες ταινίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κύριος Διακόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι προλαλήσαντες ανέφεραν πολύ σωστά επιχειρήματα. Ιδιαίτερα όταν θέλουμε να δούμε ποιες ελλείψεις και κενά υπάρχουν ακόμα σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που θα θέλαμε να αναλυθούν. Αυτά που ανέφερε ο εισηγητής είναι σωστά όλα. Σίγουρα <clears throat> θα έχουμε μια ισορροπημένη, μια ισόρροπη σωστή έκθεση ως αποτέλεσμα και όλοι θα συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια διότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα. Αλλά εκ μια παρατήρηση. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος δεν έχει ακόμα κριθεί ως προς το αν είναι καλλιτεχνική δημιουργία ή βιομηχανικό προϊόν. Αν είναι καλλιτεχνικό δημιούργημα και προϊόν πρέπει μια διαφορετική επιχειρηματολογία να υπάρξει αρχιοθέτηση των προϊόντων και τα λοιπά και αν είναι ένα βιομηχανικό προϊόν άλλα κριτήρια θα ισχύουν σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των προϊόντων. Τώρα, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή τέτοια αγορά για τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά προϊόντα, τότε θα έχουμε και τον κλασικό ανταγωνισμό στις σχέσεις μας θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τους Αμερικανούς ώστε να μην χαθεί το παιχνίδι. Αν έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν, πολιτισμικό προϊόν, μια ταινία που θα προωθείται και θα προβάλλεται σε μια διεθνή αγορά, τότε πρέπει να είναι χαμηλή η τιμή τα έξοδα ώστε να είναι ανταγωνιστικό αυτό το προϊόν με τα όσα παράγονται από πλευρά της, ε, των ΙΠΑ και άλλων χωρών. Και η ε, ρωσική αγορά είναι μεγάλη και η νότια, νοτιοαμερικανική αγορά και η βόρειοαμερικανική αμερικανικη αγορά. Γιατί να μην υπάρξει λοιπόν μια ευρωπαϊκή ε, κινηματογραφική αγορά για την διάδοση αυτών των προϊόντων. Περιορίζομαι σε αυτή την συνιστόσα. Εδώ όμως πρέπει να αποφασίσουμε, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, να αποφασίσουμε ποια συνέχεια θα δώσουμε. Και Μία ταινία παρακολούθησα που ήταν από τη Δανία ή την Σουηδία. Δεν μπόρεσα να το ε, διαχωρίσω. Την αρχή δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω. Όμως έκανα την προσπάθεια να βρω αυτή την ταινία και δεν κατάφερα να την ξαναβρω. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτά σημαίνουν ότι αυτά τα προϊόντα δεν διαχέονται στην αγορά με τον ενδεδειγμένο, τον πιο κατάλληλο τρόπο και θα πρέπει να υπάρχει και η πιστοποίηση αυτών των προϊόντων ως ευρωπαϊκών ταινιών με όλα όσα συνεπάγεται αυτό για την διάδοση και την προβολή τους. Περιορίζομαι σε αυτά τα σχόλια και θα προσπαθήσω με τον εισηγητή μέσα στο πλαίσιο σκέψεων που έχω για τροπολογίες να συνεννοηθώ μαζί. Ο συνάδελφος Τροιέσκη. Ε, Ευχαριστώ. Πάνω απ' θα ήθελα να αναδείξω τρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, η έκθεση αυτή είναι συνέχεια παλαιότερης έκθεσης. Νομίζω ο Πιότερ Μπόρις ε, ήταν ο εισηγητής τότε και νομίζω ότι ε, ε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εκείνη η δουλειά, διότι οι γνώσεις για το πώς αναπτύσσεται ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος και τι εμπόδια αντιμετωπίζει είναι πολύ κρίσιμη σημασία για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε συστάσεις στα, στους ε, εθνικούς οργανισμούς, στους εθνικούς φορείς. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα πολύ είναι η δεύτερη παρατήρησή μου, ότι θα πρέπει η έκθεση αυτή να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και οικονομικά κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο από πολλές απόψεις. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το σύστημα ε, εθνικής χρηματοδότησης ε, στην Ευρώπη ε, έχει, μεγάλες, έχει μεγάλη ποικιλομορφία. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές, υπάρχουν επιχορηγήσεις, κονδύλια και αυτό σημαίνει ότι η, διανομή των εθνικών ταινιών στην επικράτεια της Ευρώπης είναι ένα θέμα εξαιρετικά περίπλοκο γιατί δεν γνωρίζουμε πολλές φορές ποιος είναι κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε ταινίας. Και τρίτη, παρατήρηση που συζητιέται πολύ συχνά είναι η διαφήμιση, είναι η προώθηση, η εμπορική προώθηση των ταινιών αυτών. Εδώ ε, υπάρχει το, το δικαίωμα των παραγωγών να παράγουν τις ταινίες και υπάρχουν ταινίες που, ε, τα δικαιώματά τους δεν, ε, ε, που, έχουν αγοραστεί προκειμένου να μην διανομηθούν ποτέ στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για, για τέτοια φαινόμενα, συμβαίνει σε ταινίες ιστορικού περιεχομένου για παράδειγμα. Μετά, ένα άλλο ζήτημα ε, με το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξαναασχοληθεί είναι η, η μη έκδοση ταινιών. Ε, για τις ταινίες όπου δεν ήταν σαφές το καθεστώς ε, ε, ιδιοκτησίας τους, κάτι που αντιμετωπίζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα, οι μπλοκαρισμένες Και πρέπει να σας πω ότι οι μπλοκαρισμένες ταινίε υπερβαίνουν σε αριθμό τις ταινίε που παράγονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η, η αδειοδότηση, η, η, η ε, η κατανομή των δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, τα τελευταία χρόνια είχαμε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό παιδικών ταινιών. Αν όμως μιλούμε για εκπαίδευση, για παιδεία και την ε, ανάγκη να δημιουργηθεί ε, μια εκπαίδευση των παιδιών από, τα πολύ, από τις πολύ μικρές τάξεις, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολύ λίγες και κακής ποιότητας ε, παιδικές ταινίε και μάλιστα ακόμη και εκεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα στη διανομή. Και τέλος, να σας ζητήσω να θυμάστε ότι η πλειονότητα των διανομέων ε, ταινιών δεν είναι Ευρωπαίοι. Η διανομή ε, πολλές φορές βρίσκεται στα χέρια Αμερικανικών ταινιών, ε, εταιριών. Και αυτό εξηγεί εν μέρη και την ε, μεγαλύτερη προβολή αμερικανικών ταινιών παρότι η παραγωγή στην Αμερική, στις ΗΠΑ είναι μικρότερη. Οπότε θα πρέπει να καλύψουμε τρία. Ε, ε τρεις τομείς εκπαίδευση, διανομή και ε, φορολόγηση. Όλα, κολέγγε. Σαμίν και κατόπιν συνάδελφος Λιμπάτση και εδώ θα ολοκληρωθούν ε, οι παρεμβάσεις. Α, συγγνώμη, έχουμε και συνάδελφο από τη Μάλτα. Και κατόπιν θα ξαναδώσω το λόγο στο συνάδελφο Βέντα, γιατί έχουμε και την παρουσίαση της μελέτης και πρέπει να προλάβουμε και το χρόνο. Πολύ σύντομα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βέντα για την παρουσίασή του. Είναι σωστό αυτό που υπόθηκε ότι πρόκειται για συνέχιση ενός ε, θέματος που έχουμε επεξεργαστεί και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ή έχουμε τεράστιες ραγδαίες αλλαγές στο κινηματογραφικό τοπίο ε, λόγω της ψηφιοποίησης. Μιλάμε δηλαδή για την ψηφιοποίηση και των ίδιων των κινηματογραφικών αιθουσών, δηλαδή το κόστος που επομίζονται οι μικρές άθουσες και η μετάβαση από τα αναλογικά συστήματα προβολής στα ψηφιακά συστήματα είναι κάτι που ε, προκαλεί τεράστιο κόστος, πάρα πολύ μεγάλα έξοδα. Και στην Ευρώπη έχουμε πάντα το πρόβλημα ε, ότι λόγω της πολυγλωσσίας, που βεβαίως ε, από μία άποψη είναι, είναι θετικό, από την άλλη όμως για τη δημιουργία αγορών είναι πάντοτε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η αμερικανική αγορά έχει κατευθείαν 350 εκατομμύρια αγγλόφωνους ε, πελάτες συν το Ηνωμένο Βασίλειο και σύντοτι το γεγονό ότι ε, τα αγγλικά είναι μια γλώσσα ε, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένα σε όλο τον κόσμο. Αυτό βεβαίω δεν ισχύει για ταινίε που έχουν γυριστεί σε άλλε γλώσσε, πορτογαλικά, σλοβενικά για παράδειγμα. Ενώ σε αυτέ τι ταινίε πρέπει πάντοτε να, να προηγείται ο υποτιτλισμό, η μεταγλώτηση κτλ. κτλ. Και υπάρχουν και, υπάρχουν και ζητήματα συνηθιών. Στην, ε, στην ε, Γερμανία, για παράδειγμα, οι άνθρωποι περιμένουν ότι η ταινία που θα παρακολουθήσουν θα είναι μεταγλωτισμένη και όχι υποτιτλισμένη, για παράδειγμα. Είναι ε, ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα που έχει ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος έναντι του αμερικανικού. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητα καλύτερης προώθησης, καλύτερης προσβασιμότητας καλύτερης διανομής των ταινιών, ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε και πολύ μεγάλα βήματα σε αυτούς τους τομείς και στον τομέα της ψηφιοποίησης. Δεν πρέπει λοιπόν να δούμε μόνο προγράμματα προώθησης, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και την νομοθετική μας δουλειά σε μια σειρά από εμπορικούς τομείς. Είναι σωστό. Ε, πολλές φορές ε, ε, μπλοκάρουμε ε, εμείς οι ίδιοι του ε, παρόχους μας και μετά έρχεται για παράδειγμα το, το, το Netflix και επειδή είναι αμερικανική εταιρεία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, θα πρέπει εμεί νομίζω από νομοθετική πλευρά δηλαδή να αναλάβουμε κίνηση τι ώστε να, διο, να, να διευκολύνουμε την διανομή των ευρωπαϊκών ταινιών. Υπάρχουν και τα blockbuster, υπάρχουν όμως και γερμανικές και γαλλικές ταινίες που νομίζω ότι έχουν, ε, είχαν και μεγάλη διεθνή κοινή απήχηση. Υπήρχαν και τα τελευταία χρόνια και Ιταλικέ ταινίε οι οποίε έγιναν ευρύτατα γνωστέ σε όλο τον κόσμο. Αλλά πράγματι είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ο Ευρωπαϊκό ε, κινηματογράφος μένει εγκλωβισμένο σε αυτές τις μικρές ε, ε, ε, αίθουσες και δεν καταφέρνει να φτάσει στις μεγάλες αίθουσε προβολής. Αυτό οφείλεται και στη διαφήμιση και σε δομικά προβλήματα. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να απλοποιηθεί και το σύστημα των πνευματικών δικαιωμάτων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα του, περιεχομένου αλλά ε, θα πρέπει στο μέλλον να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότηση ε, για όλη την αλυσίδα αξίας, όχι μόνο για την παραγωγή της ταινίας, αλλά για όλα τα στάδια. Και στην αναδιάρθρωση αυτών των δομών που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τόσο την ελκυστικότητα των κινηματογραφικών αιθουσών, αλλά να ιχνηλατήσουμε και νέες μεθόδους διανομής των ταινιών, DVD, video on demand, πέραν της παραδοσιακής οδού, της τηλεόρασης δηλαδή. Γιατί υπάρχουν και διαφορετικές απαιτήσεις πλέον από την πλευρά των χρηστών. Οι χρήστες σήμερα μετά την, κινηματογραφική, την έναρξη της κινηματογραφικής προβολής θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ταινία και αυτό πολλές φορές για νομικούς λόγους δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Φυσικά αυτό αφορά και τις κινηματογραφικές αίθουσες γιατί αν ε, οι ταινίες διατίθενται online λίγο μετά το λανσάνισμά τους στην κινηματογραφική αίθουσα οι άνθρωποι θα κάτσουν στα σπίτια τους που έχουν πλέον και αυτές τις μεγάλες οθόνες και, και, είναι αλήθεια ότι αυτή η αίσθηση και αυτή η νέα τεχνολογική δυνατότητα να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ταινίες στο σπίτι του σαν να βρίσκεται σε κινηματογράφο θα, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις κινηματογραφικές αίθουσες. Όπως είπαμε, ε, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, υπάρχουν πάρα πολλές πολιτισμικές ε, πτυχές αλλά θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας και να μπορέσουμε να τα εξυπηρετήσουμε και ελπίζω στην ε, έκθεση να μην αναδείξουμε μόνο τα πολλά επίπεδα των προβλημάτων, αλλά ότι θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και συγκεκριμένες λύσεις για το πώ θα μπορέσουμε να δώσουμε στο μέλλον απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ Σαμπίνα. Και τώρα συνάδελφο από τη Μάλτα Πολυμπάτσικα. Θα ήθελα να πω πολύ ειλικρινά ότι ένα από τα προβλήματα του Ευρωπαϊκού είμαστε εμεί. Δηλαδή το βάρο που έχει η πολιτική στι επιλογέ και είναι μια πολιτική που κάνει επιλογέ ε, βάσει πολύ μικρών ικανοτήτων. Και υπάρχουν όμως και κάποια πολύ καλά παραδείγματα. Το γαλλικό σινεμά, παραδείγματος χάρη, είχαμε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, κυρίως στην περίοδο όταν ήταν ε, η Λαγκάρε υπουργό πολιτισμού, ε, πρόθυσε πολύ το γαλλικό αυτό κλάδο και είναι τώρα και υψηλή ποιότητα. Και είχαμε και στην Ιταλία ε, κάποια σημαντικέ ταινίε. Έχουμε σήμερα στην Ιταλία μια ταινία του φίλου μου Μάριο Ματώνε που αφορά έναν ποιητή ε, του 1800, τον Τζέκομο Λεοπάρντι και έχουμε πάρα πολύ ψηλά εισιτήρια σε αυτή την ταινία και ε, η διαφορά με την ταινία του Μαριο Μερτώνε ε, είναι ότι υποστηρίχθηκε από το κράτος η διανομή της ταινία. Υπήρξε και ένας νόμος που επέτρεψε να υπάρξει καλύτερη συγκέντρωση ιδιωτικών κονδυλίων ε, για να δημιουργηθεί αυτή η ταινία που ήταν και δαπανηρή και αυτό λειτουργήσε. Έτσι λοιπόν για μια φορά η πολιτική έκανε μια σωστή επιλογή υποστήριξης και πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Πολύ συχνά όμως η πολιτική κάνει κάποιες επιλογές οποίε είναι μεροληπτικέ ή δεν βασίζονται σε επαρκή γνώση. Εγώ ειλικρινά θέλω να πω το εξή. Εγώ είμαι καινούριο εδώ και μιλώ λίγο. Ακούω του πιο πειραμένου συναδέλφου. Όμω και σήμερα το πρωί άκουσα κάποια παράδοξα θέματα. Ε, υπήρξε και μία πολεμική για το ότι ποτέ δεν κέρδισε το βραβείο Λουξ μία ε, κομμωδία. Πριν από κάποια χρόνια ε, κέρδισαν τα χιόνια του Χιλιμάντζερο, που δεν είναι κομμωδία, αλλά ήταν μια πολύ αστεία ταινία, με τις πιο αστείες που έχω εγώ δει. Και ε, πιο πριν υπήρξε και μία συζήτηση για μία σειρά εμπειρογνωμόνων που πρέπει να ακούσουμε σε σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά. Εγώ, συγγνώμη τώρα που τα λέω, αλλά δεν μπόρεσα ε, να μιλήσω προηγουμένως. Είχαμε έναν εμπειρογνώμονα για τα πολιτιστικά αγαθά που έχει αναγνωριστεί ω τέτοιο από όλους τους διεθνεί οργανισμούς, από τι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Γερμανία, το Σαλβατόρε Σέτι και πιθανότητα ε, γιατί προτάθηκε από μια πιο μικρή πολιτική ομάδα και προτιμήθηκαν εμπειρογνώμονες που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ και δεν έχουν δημοσιεύσει ποτέ ούτε καν ένα βιβλίο για τα πολιτιστικά αγαθά στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν οι επιλογές των πολιτικών στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και συγκεκριμένα των κινηματογράφων όπου δεν έχουμε στη διάθεσή μας μεγάλα κεφάλαια όπως ισχύει στη Μεγάλη Βορειοαμερικανική αγορά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε μια αυτοκριτική του ρόλου της πολιτικής στην προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας και του κινηματογράφου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ συνάδελφε και τώρα θα δώσω το λόγο ε, συνάδελφο Λιμπάτσκα και κατόπιν θα ήθελα να ρωτήσω από την Κομισιόν αν θέλει κάποιο να πάρει το λόγο πριν να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Έχουμε εκπροσώπους από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Connect, την Λαγκάρη, Καρολίλα Λεφλερότ. Θα ήθελα να τους ρωτήσω αν κάποιος από αυτούς θα ήθελε να πάρει το λόγο. Διαφορετικά θα κλείσουμε με τον συνάδελφο Βέντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βέντα που προετοίμασε αυτή την γνωμοδότηση. Η συζήτηση που είχαμε για τον κινηματογράφο στην Ευρώπη έναντι του Αμερικανικού κινηματογράφου είναι πραγματικά μια συζήτηση που αφορά κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλουμε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός να συνεχίσει να είναι ένας πολιτισμός που θα αντικατοπτρίζει την πολιτιστική μας ε, κληρονομιά ή θέλουμε τελικά ένα πολιτισμό ε, που θα είναι γελίος, κάτι που βλέπουμε σε πολλές αμερικανικές ταινίες. Αν ε, μιλάμε για αυτή ε, τη δυσανάλογη σχέση μεταξύ της Αμερικανικής αγοράς ε, και της Ευρωπαϊκής αγοράς, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να προσθέσουμε και πολλά άλλα πρότυπα ως τεράστια διαφορά, γιατί αυτές οι αγορές είναι κατακαιρματισμένες. Εμείς ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία κυρία σημεία που θα πρέπει να αναπτύξουμε συστηματικά. Καταρχήν, να καλλιεργήσουμε ε, στους θεατές ε, μια κουλτούρα να θέλουν να παρακολουθούν ποιοτικά ε, ποιοτικές ταινίε ε, και όχι βίαιες ή γελίες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. Δεύτερον, θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε το σύστημα της διανομής, επειδή έχουμε τεράστια ανάπτυξη της ψηφιακή αγοράς. Τρίτον, και εδώ συμφωνώ με την Πρόεδρο, όταν μιλάμε για την ανάγκη της δημιουργίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ναι, ναι, συμφωνώ. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά που θα σε χρηματοδοτεί τα project και θα διατηρήσει και την πολυπλωσία στον κινηματογράφο. Και φυσικά συμπεριλαμβανομένου και του υποτιτλισμού και του dubbing. Όμως πρέπει να δούμε και την ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ τη αγγλικής γλώσσα και των άλλων γλωσσών. Και όπως σας είπα αυτό αφορά όλο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όχι μόνο τον κινηματογράφο. Και φυσικά πρέπει να δούμε και ποια είναι και η ιστορική πηγή του διαφωτισμό. Υπάρχουν παρεμβάσει από την πλευρά τη Κομισιόν. Όχι. Μάλιστα. Α, με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Κύριος Λαγκάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας ε, και τον κύριο Βέντα για την υποστήριξή του, κυρίως ό,τι αφορά την οργάνωση του φόρουμ για τις ταινίε. Η Κομισιόν έχει δει τοποθετηθεί στην ανακοίνωση της ε, σαφέστατα, οπότε δεν θα επανέλθω σε αυτά τα αυτά. Αποτελεί μια ανάλυση του οπτικοακουστικού κλάδου και αναφέρεται και στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κλάδος αυτός, κυρίως στα πλαίσια της ψηφιακής επανάστασης. Όπως αναφέρθηκε ήδη από πολλούς ομιλητές, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα, γιατί ε, περιλαμβάνει και ρυθμιστικές πτυχές και πτυχές χρηματοδότησης και πτυχές εκπαίδευσης ε, αλλά και πάρα πολλούς παράγοντες που παρεμβαίνουν. Και γι' αυτό η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της ε, ήθελε να δημιουργηθεί αυτό το φόρουμ για τις ταινίε έτσι ώστε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν και όσοι δραστηριοποιούνται στον οπτικοφυστικό τομέα αλλά και όσοι δραστηριοποιούνται και πέραν αυτού. Και είχαμε κατά νου κάποιες εταιρείες όπως τη Netflix, κάποιες νέες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, αλλά φυσικά θέλαμε να βάλουμε και το κοινό σε αυτό το παιχνίδι. Προς η μορφή ε, αυτών των συγκεκριμένων ταινιών και το φορμά τους είναι υπό εξέταση. Απριόρι θα πρέπει να βασιστούμε σε εφιστάμενα μέσα και παρέχονται ήδη από το πρόγραμμα Media. Για να ολοκληρώσω, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει πραγματική βούληση να βράξουμε τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί από αυτή την ανακοίνωση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα διαρθρωμένο διάλογο για αυτή τη θεματική. Και φυσικά και το Κοινοβούλιο με την εμπειρία του και την υποστήριξή του θα είναι ένας μεγάλος παίκτη σε όλη αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Βέντα, θέλετε να ολοκληρώσετε, παρακαλώ. E, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω όλους για τα ερωτήματα και τις παρεμβάσεις τους και για τις προτάσεις τους. Ζήτησα βοήθεια και Επαναλαμβάνω το αίτημα αυτό και ευχαριστώ για την δυνατότητα αυτών των προτάσεων. Και ίσως τώρα μια και έφυγε η Πέτρα. Αυτό το οποίο ανέφερε για τις δύο όψεις του νομίσματος, την οικονομική ή την μία όψη και την άλλη την πολιτισμική ή την καλλιτεχνική. Και για την εμβέλεια είναι δύσκολο καμιά φορά να διαφοροποιήσει κανείς ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των επιλογών. Η αλυσίδα της διανομής πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί, διότι οι άλλες δυνατότητες διάθεσης, για παράδειγμα βίντεο και σύναφων προϊόντων, είναι κάτι το κατάλληλο να μπορέσουμε να συναγάγουμε συμπεράσματα, να μάθουμε και να δράσουμε αντίστοιχα και προς εμάς ευχαριστώ για την πρότασή σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό το οποίο διανοίγεται εδώ. Και βασιζόμενος σε σχέση με τη, τα στοιχεία του Επιτρόπου Oettinger που προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν και αναφέρθηκαν για το τι χρειαζόμαστε σε σχέση με το μέλλον ώστε να μπορέσουμε καινοτόμα προϊόντα να δημιουργήσουμε σε σχέση με το πλαίσιο για την προστασία πνευματικών ε, δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παραγωγού, copyright στην ψηφιακή εποχή, θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, θέματα που απασχόλησαν και τον Επίτροπο και για την συμμετοχή από πλευράς μας σε συγκεκριμένες συναντήσεις ε, με εμπλεκόμενους και εκπροσώπους των διαφορών τομέων και του οπτικοακουστικού τομέα για, το οποίο, αυτό, για τον οποίο τομέα είναι πολύ σημαντικά τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και ποιες λύσεις πρέπει να στοχεύσουμε στο μέλλον να υιοθετηθούν. Θα το ξαναδούμε και θα επιστρέψουμε σε αυτό και θέλω να ευχαριστήσω για την αναφορά αυτή από πλευρά σας. Τώρα δεν βλέπω την Σάντι που θα μπορούσα να απαντήσω ότι πρόκειται εδώ για αυτό, για υποτιτλισμούς, υποτιτλισμούς σε ταινίε. Βρισκόμαστε στο εξωτερικό για παράδειγμα και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια ταινία χωρίς υποτιτλισμό όπως αναφέρθηκε και από τους σκιώδεις εισηγητές, από σκιώδη εισηγητή. Σίγουρα Πολλές φορές στη σταδιοδρομία μου το παρατήρησα και με τα βιώματά μου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Υπήρχε μια ενδιαφέρουσα ταινία που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω επειδή δεν μπορούσα να την ε, παρακολουθήσω ή να την βρω από πλευράς γλωσσικής ε, κατανοητή. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε πώς μπορεί να επιληθεί. Ένα τρόπο χωρίς ε, ε, συνδρομή ή τέλη για τους ε, νέους χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος για παράδειγμα να μπορούν να κατεβάζουν τέτοια προϊόντα σε, στην εποχή την διαδικτυακή, διαδικτυακά προϊόντα και να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο νεότερος αυτό, η, ο τομέας αυτός των νεότερων θεατών περισσότερο. Αυτά σε σχέση με την απουσία του συναδέφου και εδώ συνεχίζω σε σχέση με τον αξιότιμο συνάδελφο που απουσίασε. Θα θέλω όμως να αναφέρω σε σχέση με αυτό το θέμα ότι διαδικτυακά οι θεατές ή για το ζήτημα αν μπορεί το θέμα των, ε, της πολιτιστικής αξίας τέτοιων προϊόντων και αν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν ε, προϊόντα των είπα, Είναι ένα πραγματικά σημαντικό θέμα και ευχαριστώ για το ότι μου δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθώ. Υπάρχουν δύο θέματα για την διανομή και την ε, ε, αγορά. Αν έχουμε ένα ρουμανικό προϊόν, πολωνικό ε, και για την αδειοδότησή του ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση σχετικά γιατί αν δεν το κάνουμε δεν θα έχουμε καμιά ευκαιρία να ανταγωνιστούμε ισχυρούς, ε, ισχυρούς ομίλους ε, διανομής ε, και αυξανόμενη ζήτηση ευρωπαϊκών ταινιών. Ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη. Τέχνη τώρα, καλλιτεχνική συνιστόσα για αυτή την παρέμβαση αν είναι καλλιτεχνικό προϊόν ή βιομηχανικό προϊόν μια ταινία. Υπάρχουν πολλά συνεμπλεκόμενα θέματα εδώ και πρέπει να δούμε και το ίδιο το θέμα της πλατφόρμας, ενός πυλώνα που θα υποστηρίζει τέτοια προϊόντα είναι ένα ευρύτερο ζήτημα και θα πρέπει να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να απαντηθεί μέσα από την έκθεσή μου. Ελπίζω από κοινού μαζί σας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία επ' αυτού και πιστεύω στα γερμανικά. Ψηφιακή εποχή, κόστος όσον αφορά αυτά τα προϊόντα της ταινία, όπως ανέφερα στην έκθεσή μου και εγώ Είμαι συνεφίλ, είμαι ιδιαίτερα θερμός οπαδός των ταινιών. Το να μπορέσει κανείς να δει μια ταινία κατεβάζοντάς την δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος. Δεν είναι το ίδιο με το να παρακολουθήσει κανείς μια ταινία στην κινηματογραφική οθόνη, στον κινηματογράφο, σε ένα περιβάλλον με ε, φίλους ε, είναι πολυσχηδής ο κόσμος μας και μεταβάλλονται όλα με ραχδαίους, με ταχύς ρυθμούς. Και φυσικά στη διεθνή αγορά χρειαζόμαστε νέες δομές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Η εξέβρεση αυτών των δυνατοτήτων λοιπόν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε βελτιωμένη πρόσβαση στους χρήστες, σε όλους εκείνους που πραγματικά ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα προϊόντα και την ε, το να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες για τις ταινίε καλύτερα. Μια στιγμή. Ε, μπορώ να συνεχίσω. Πολωνικά θα είναι πιο εύκολο να μπορέσω να τοποθετηθώ. Σε σχέση με το βίωμα αυτό βλέπουμε ότι σήμερα γίνονται σχετικές έρευνες για το οικονομικό, την οικονομική συνιστόσα για τις επιχορηγήσεις και τις επιδοτήσεις ουσιαστικά υπάρχει και η συνιστόσα του να αγοράζονται τα δικαιώματα μιας ταινίας και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές εκμετάλλευσης αυτής της ταινίας ή ποιες δεν θα είναι το τι γίνεται σε σχέση με το Κοινοβούλιο για το πώς θέλουμε να προστατεύσουμε ε, τις ταινίε από το να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, σε έναν μονόδρομο. Ναι, ολοκληρώνω και για τον συνάδελφο για την παρατήρηση που έκανε η, η διανομή που δεν είναι σήμερα ευρωπαϊκή. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια και συμφωνούμε για την συνεισφορά που μπορεί να υπάρξει. Σας ευχαριστώ και σημειώνω αυτή την παρέμβασή σας που θα λάβω ιδιαίτερα υπόψη για την διανομή των ταινιών και σε σχέση με την εκπαίδευση για να δημιουργηθεί η πλατφόρμα εκείνη θεατών που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ συνάδελφε Βέντα. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα θέμα που ενδιαφέρε όλους τους συναδέλφους. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή την ισορροπία που πρέπει να εγγυηθούμε για να αναπτύξουμε και το κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή. Ο κινηματογράφος ε, είναι και βιομηχανία αλλά και δημιουργικότητα και τα νέα μέσα θα μας επιτρέψουν να υποστηρίξουμε περισσότερο τη διανομή, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και μια σειρά αξίας έτσι ώστε και η ίδια η παραγωγή να έχει την δυνατότητα να επενδύσει. Φυσικά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και το νέο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe, έχει δώσει μεγάλη έμφαση στο θέμα της διανομής, όμως τα προβλήματα είναι αυτά που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Έτσι λοιπόν, η προθεσμία για την παρουσίαση της έκθεσης είναι τον Ιανουάριο και θα ψηφίσουμε τον Μάρτιο. Θα ήθελα τώρα, πολύ σύντομα, να σας πω για τους συντονιστές. Είχαμε μία συνεδρίαση συντονιστών με πάρα πολλά ζητήματα που έπρεπε να αποφασίσουμε. Δεν εξαντλήσαμε όλα τα θέματα και έτσι Λοιπόν, θα συζητηθούν ε, τα τελευταία θέματα που μας έμειναν σε μια επόμενη συνάντηση, όμως να σας ενημερώσω για το τι αποφασίστηκε. Αποφασίστηκε να προδιατεθούν κάποιες ε, γνωμοδοτήσεις σε ό,τι αφορά την πνευματική διοκτησία, το copyright ε, και θα είναι η ομάδα των πρασίνων που θα την αναλάβει. Μια άλλη έκθεση για την οικονομική, και κοινωνική, εδαφική συνοχή που σχετίζεται με την Επιτροπή Ρέτζη. Θα είναι δική μου αρμοδιότητα γιατί δεν υπήρχαν ομάδε που έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον. Νομίζω όμω ότι η Επιτροπή πρέπει να τοποθετηθεί για ένα τέτοιο θέμα. Θα έχουμε και μία έκθεση που θα ανατεθεί στους φιλελεύθερους για την πράσινη βίβλο, για ε, οι γεωγραφικέ ενδείξει και για την προστασία για τα αγροτικά προϊόντα, για την ημικό. Σε ό,τι αφορά τώρα Άλλο θέμα, ζητήσαμε από τη Γραμματεία να λάβει συγκεκριμένε πληροφορίε για δύο θέματα. Για το στάδιο εφαρμογή τη οδηγία για το Collecting Societies και για τα δικαιώματα δημιουργού, για τη μουσική. Και ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να εμβαθύνουμε έχει να κάνει με ένα αίτημα που είχε να κάνει με τα τέλη πιστοποίησης που φαίνονται να πληρώνουν στο ραδιόφωνο κάποια αθλητικογράφοι σε ορισμένες χώρες. Σε ό,τι αφορά το European Heritage Label που είναι το νέο πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν, δια, πριν δύο χρόνια και είναι σε στάδιο εφαρμογής, αποφασίστηκε να ε, επιβεβαιώσουμε την επόμενη περίοδο, να επαναδιορίσουμε τους τέσσερις ε, εμπειρογνώμονες, γιατί αναγνωρίζαμε την αξία τους, αλλά θεωρούμε ότι είναι και σημαντικό να προσπαθήσουμε να δώσουμε μία συνέχεια σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και γι' αυτό εγώ θα σας πρότεινα τον Ιανουάριο Ίσως να καλέσουμε αυτούς τους εμπειρογνώμονες για μια ακρόαση για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πρόγραμμα. Ένα άλλο σημείο. Ε, Επιβεβαίωσαμε το ενδιαφέρον της Επιτροπής μας ε, να διοργανώσει μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή ΕΜΠΛΕ για τα επικαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη ως τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, ως μια οδό κατά πολέμηση ενεργείας των νέων το πρώτο εξάμεινο του 2015 και κατόπιν εντοπίσαμε και τους εμπειρογνώμονες για την ακρόαση για την πολιτιστική κληρονομιά και αναφέρομαι και στο συνάδελφο Μαλτέζα. Υπήρξε μία δύσκολη συμφωνία μεταξύ των συντονιστών θα έχουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες και δύο αναπληρωτές τον καθηγητή Πούρτσλα, την κυρία Μπενεντίτ Σέφλανξ, τον σοσιαλιστό αρχιτέκτονα και τον καθηγητή Τζόνς. Και οι αναπληρωτές θα είναι ο δόκτωρ Κάρλο Μινέλη και η δόκτωρ Τερέζα Μινέλη. Τέλα, να συγχωρείτε. Αυτά σε σχέση με τις αποφάσεις των συντονιστών. Και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην παρουσίαση της μελέτης ε, του θεματικού τμήματος Β για τους τίτλους για την εισαγωγή και την ενότητα εκπαίδευση εξετάσεις στην Ευρώπη. Μια συγκριτική μελέτη, μια ενδιαφέρουσα συγκριτική μελέτη. Εδώ έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικολό Ντουράτσι από το LCE Enterprise και την κυρία Σεσίλ Παρό, Μαγκράθ από το Rand Europe. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας γιατί αφορά ακριβώς την ευκαιρία μιας πραγματικής ε, κυκλοφορίας και κινητικότητας ε, για την ανώτητη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Ενδιαφέρει αυτό και τους νέους αλλά και τους ε, ενήλικες γιατί μια τέτοια σύγκριση θα μπορούσε να αποτελέσει και μια βάση να συζητήσουμε και να βαθύνουμε στο θέμα ως Επιτροπή Πολιτισμού. Για να μην χάνουμε χρόνο, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Όνομα μου είναι Νικόλο Ντουράτσι. Είμαι εδώ με την συνάδελφό μου Σεσίλ Χορό από τη Rand Europe Γνωρίζουμε του ε, χρονικού περιορισμού, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται. Είμαστε εδώ για να σα παρουσιάσουμε μια μελέτη που διεξήχθη μεταξύ Ιουλίου 2013 και Μαρτίου 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε από το LSE Enterprise και τη RAND Europe. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ε, η μελέτη αυτή γιατί εξέτασε τα συστήματα εισαγωγή στην Ευρώπη και πέραν από την Ευρώπη και θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω σε λίγα λεπτά τα πορίσματα της έρευνας, της μελέτης αυτής και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να εξετάσουμε ενδεχομένως και τα, τα λεπτομεριακά στοιχεία που αφορούν αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, η δομή της παρουσίασης είναι απλή. Έχουμε τρει, τρεις ε, βασικούς τίτλους. Η Σεσίλ θα περιγράψει το τοπίο ε, εισαγωγικά εγώ στη συνέχεια θα σας δώσω μια σύνοψη των βασικών πορισμάτων που προέκυψαν από την έρευνα αυτή και στη συνέχεια θα ξαναδώσω το λόγο στη Σεσίλ για να διατρέξει τις συστάσεις πολιτικής ε, στις οποίες καταλέξαμε. Μια σειρά από πρωτοβουλίες που ενδεχομένως δηλαδή θα είχαν ε, ενδιαφέρον να τα εξετάσουν τα θεσμικά ε, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, οπότε δίνω το λόγο τώρα στη Σεσίλ. Ευχαριστώ Νικολό και ευχαριστώ που μας καλέσατε σήμερα, κυρία Πρόεδρε, ε, μέλη της Επιτροπής. Ε, και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το γεγονός βεβαίως ότι μας δόθηκε ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό το συναρπαστικό θέμα. Λοιπόν, το υπόβαθρο της, ε, μελέτης. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια πρόκληση. Αφενός έχουμε ε, μια ε, πρόκληση να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες δεξιότητες. Από την άλλη πλευρά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν περιορισμούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο αυξανόμενο αριθμό φοιτητών. Για παράδειγμα, έχει ε, αυξηθεί κατά 25% μεταξύ 2005 και 2005 ο αριθμός των νέων εισερχομένων. Αλλά ταυτόχρονα ε, τα ιδρύματα ε, έχουν να αντιμετωπίσουν μειωμένους προϋπολογισμούς. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε βοηθήσουμε τα Ιδρύματα ώστε να ανταποκριθούν. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη να, ε, να υπάρξει μια ρύθμιση του, του, ε, του αριθμού των ε, ε, ε Υπάρχει ανάγκη να αντιστοιχηθούν οι φοιτητές στις, στους κύκλους σπουδών και τα συστήματα εισαγωγή μπορούν να βοηθήσουν στο να επιλεγούν οι καλύτεροι φοιτητέ για να βελτιωθεί και η ποιότητα της ανώτατη εκπαίδευση. Εκτός λοιπόν από... Εξετάσαμε λοιπόν τόσο τα συστήματα εισαγωγής όσο και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή. Από, το τέλος της δεκαετίας 90 λοιπόν έχουν υπάρξει πάρα πολλές ε, μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας Μπολόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο το ενδιαφέρον δεν ήταν ε, ε, το απαραίτητο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και σε πάρα πολλές χώρες υπάρχουν ακόμα τυπικές και πολύ στέρεες ε, διαδικασίες για την εισαγωγή. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τα συστήματα αυτά έχουν παραμείνει εν πολλής η ίδια, υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς εξελίξεις που είναι ραγδαίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί ε, νέοι διεθνείς φοιτητέ. Μεταξύ 2005 και 2011 αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο οι φοιτητέ που εισέρχονται από, το, από, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πανεπιστήμια μας. Γι' αυτό πρέπει πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή όσον αφορά την αναγνώριση. Επίσης υπάρχει και ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό ε, περιβάλλον. Υπάρχουν ε, νέες δυνατότητες όπως για παράδειγμα τα ψυχομετρικά δεδομένα που ανοίγουν το δρόμο για να κάνουμε ακόμα καλύτερες δοκιμασίες ε, καταλληλότητας. Η τεχνολογία θα μπορούσε να μας βοηθήσει και στο πώς διαχειριζόμαστε τις αιτήσει. Παρά τις, γεγονο... τις αλλαγές αυτές όμως, οι βασικοί δείκτες δείχνουν ότι τα συστήματα εισαγωγής δεν κάνουν ό,τι θα μπορούσαν, το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν. Και εδώ βλέπετε ε, ότι τα ποσοστά αποφύτησης διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο 50% ε, θα αποφυτίσει των φοιτητών αυτός ο αριθμός μειώνεται στο 1 τρίτο σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γερμανία. Αυτό μας ανησυχεί γιατί βασικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι ε, πολλά συστήματα τελικά καταλήγουν σε αποτυχία των φοιτητών και αυτό είναι ανησυχητικό διότι, οι χώρες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό νεοεισερχομένων δεν είναι εκείνες που έχουν τους περισσότερους αποφύτους και εδώ μπορείτε να δείτε διαφορά μεταξύ των ποσοστών εισαγωγής και των ποσοστών αποφύτου συζήτηση, για παράδειγμα σε χώρες όπως η Σλοβονία. Θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσετε το κεφάλαιο 1 αν θέλετε να, έχετε, αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Το υπόβαθρο στη συνέχεια ε, είναι το εξής. Για ποιο λόγο έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό φοιτητών και παρότι δεν λέμε ότι τα συστήματα εισαγωγής μπορούν να λύσουν όλα μας τα προβλήματα στην ανώτερη εκπαίδευση, παρόλα αυτά φαίνεται ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν συστήματα εισαγωγής τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τη ρύθμιση των ποσοστών εισαγωγής και αποφύτησης. Και τα απορρίσματα μας δείχνουν ότι τα συστήματα εισαγωγής είναι λειτουργικά αν ανταποκρίνονται σε τρία κριτήρια. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ισότητα. Δεν θα πρέπει δηλαδή μόνο να αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις των, ε, ε των ετούντων, αλλά θα πρέπει να βοηθούν και στους φοιτητές να επιτυχάνουν ε, τα καλύτερα αποτελέσματα στη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης θα πρέπει τα συστήματα εισαγωγής να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθούν τους φοιτητές να είναι οικονομικά βιώσιμα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για τις εθνικές διοικήσεις. Και τέλος τα συστήματα εισαγωγής θα πρέπει να διασφαλίζουν την κινητικότητα των φοιτητών. Αν θέλουμε να ε, επιτύχουμε τον στόχο για 20% ε, κινητικότητα στους φοιτητές. Η ε, μελέτη απάντησε τρία ε, ερωτήματα. Πώς μπορούν τα συστήματα εισαγωγής να βοηθήσουν την κινητικότητα των φοιτητών. Δεύτερον, πώς μπορούν αυτά τα συστήματα, πώς αυτά τα συστήματα προωθούν την, την κινητικότητα και την ποιότητα και την ισότητα των ε, φοιτητών. Τα τρία ερωτήματα αυτά ε, είναι σημαντικά για το αν θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση σε ενωσιακό επίπεδο. Ε, όλα αυτά τα ερωτήματα μπορούν να συγχωνευτούν σε, σε ένα ερώτημα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν τις διαδικασίες τους και ε, διεξήγαμε στη βάση αυτή μια συγκριτική μελέτη 10 χωρών ε, ευρωπαϊκών αλλά και χωρών από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, επιλέξαμε τις χώρες αυτές ακριβώς γιατί αντιπροσωπεύουν ένα μείγμα συστημάτων εισαγωγής. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα, για προσόντα που αποκτήθηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη Γαλλία είναι το μπακαλωρεά, στη Σλοβενία είναι το ματσού και συγκρίνουμε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες με τις ξένες χώρες στη βάση ε, του πόσο γνωστά είναι τα συστήματά τους. Για παράδειγμα υπάρχει το αμερικανικό σύστημα όπου υπάρχουν τα τυποποιημένα ε, τεστ που έχουν ορισμένες, που έχει η Αυστραλία για παράδειγμα έχει ένα σύστημα με πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές και έχουμε και την Τουρκία και την Ιαπωνία λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στην ε, Ιαπωνία και την Τουρκία την χρησιμοποίησαμε ως γειτονική χώρα. Ο συνάδελφός μου θα σας δώσει ε, μια σύνοψη των βασικών πορισμάτων ε, όσον αφορά αυτές τις τρεις, τους τρεις άξονες της ισότητας, της κινητικότητας και της ποιότητας. Λοιπόν, το ζήτημα της ισότητας βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και θα χρειαζόταν πάρα πολλής χρόνος για να σας το περιγράψω σε βάθος. Αλλά για να σας πω το, τα βασικά, τα θεμελιώδη στοιχεία. Αυτό που κάναμε ήταν ε, ε, ότι παρήχαμε κάποιες ε, πληροφορίες για τα συστήματα εισαγωγής των χωρών, ανοιχτή πρόσβαση, επιλεκτική πρόσβαση και πώς αυτά τα συστήματα αποδίδουν, τι αποτελέσματα αποφέρουν στην, στα, στα, όσον αφορά την ισότητα και την ποιότητα. Λοιπόν, ε, όσον αφορά την ποιότητα και την πρόσβασιμότητα της ε, ανώτατης εκπαίδευσης, αυτή συνήθως μετράται στο... Ε, ε, ε βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο, το αν δηλαδή θα πάρω πτυχίο βασίζεται και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους γονείς μου. Ε, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στα συστήματα λοιπόν αυτά. Και αυτό που βλέπουμε είναι, ε, είναι κάπως ανησυχητικό ή κάπως παραπλανητικό. Δεν βλέπουμε συσχετισμό με τον, ε, ανάμεσα στις χώρες που επιτυχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα συστήματα εισαγωγής τους. Οι χώρες που έχουν ή η ίση, για παράδειγμα, αποτελεσματικότητα, βλέπετε εδώ Σλοβενία, Φιλανδία, έχουν και ανοιχτά και κλειστά συστήματα, επιλακτικά συστήματα εισαγωγή. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, στη Γερμανία ότι υπάρχει ένα ανοιχτό σύστημα επιλογή. Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι, λοιπόν, ότι ο συσχετισμό μεταξύ μια τυπολογία ε, συστημάτων εισαγωγή και των επιδόσεων που έχει το σύστημα αυτό όσον αφορά την ποιότητα είναι πολύ περίπλοκος τα, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία τα συστήματα εισαγωγή μπορούν να τα κάνουν και κάποια που δεν μπορούν να κάνουν. Ποια είναι λοιπόν τα πράγματα που μπορούν να κάνουν, τι που δεν, δεν μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν τα συστήματα εισαγωγή. Δεν μπορούν να ε, αντιμετωπίσουμε φυσικά το ζήτημα των τριών αξώνων που περιέγραψα μέσω του συστήματο εισαγωγή. Να σα δώσω ένα ε, παράδειγμα. Υπάρχουν ε, παραδείγματα χωρών όπου ε, όπου οι μαθητές πολύ νωρίς, οι μαθητές και φοιτητές πολύ νωρίς μπαίνουν σε καλούπια εκπαιδευτικά. Ε, είναι σαφές σε αυτές τις περιπτώσεις ε, ότι το σύστημα εισαγωγής τους επηρεάζει διότι γιατί το αν θα μπουν στο πανεπιστήμιο ή όχι αποφασίζεται πολύ νωρίς. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε να, να εξετάσουμε το ζήτημα της ισότητας και της ποιότητας μόνο μέσω των συστημάτων εισαγωγής. Και πράγματι η ανοιχτή πρόσβαση δεν συνεπάγεται απαραίτητο τουλάχιστον ότι το σύστημα ανώτητη εκπαίδευση θα είναι και πιο ίσο, θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ισότητα. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια πράγματα που τα συστήματα εισαγωγή μπορούν να κάνουν για να καταστήσουν την ε, ε περισσότερο ισότιμη την ανώτητη εκπαίδευση. Και εδώ θέλω να τονίσω κάτι ε, που προκύπτει και από τις συνεντεύξεις με τους ενδιαφερομένους, ότι τα συστήματα εισαγωγής δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στη διαχείριση της πρόσβασης, αλλά θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι φοιτητέ θα ολοκληρώνουν τους κύκλους σπουδών τους. Και αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητέ θα πρέπει να έχουν όσο το περισσότερες δυνατόν, όσο το, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο. Και να διασφαλίζουμε ότι ο κύκλος σπουδών που επιλέγουν είναι ο κατάλληλος για εκείνους, ώστε να διασφαλίσουμε και την πιθανότητα να αποφυτίσουν στο τέλος. Υπάρχει λοιπόν μια πτυχή ισότητας και πτυχή ποιότητας σε αυτό το θέμα. Ε, φυσικά η αύξηση του ποσοστού αποφυτισής είναι σημαντικό, αλλά η αύξηση του ποσοστού αυτού μέσω της παροχής πληροφοριών πριν από την εγγραφή τους είναι και ένας ε, άξονας ισότητας, διότι γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που έχουν λιγότερη πρόσβαση στην πληροφορία είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις ε, λιγότερο ενημερωμένες επιλογές και λαμβάνουν τις, τις χειρότερες αποφάσεις συγκριτικά. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των συστημάτων εισαγωγή και την προσβασιμότητα στην ανώτερη εκπαίδευση. Δύο θέματα. Αν κάποιο θέλει να εξετάσει με σοβαρού όρου τη διεύρυνση τη πρόσβαση στην ε, ανώτερη εκπαίδευση, θα πρέπει να εξετάσει και τα συστήματα εισαγωγή και τα συστήματα εισαγωγή να δίνουν όσο το περισσότερο πληροφορίε γίνεται στου ετούντε, προκειμένου να μην μπαίνουν μόνο οι φοιτητέ στα πανεπιστήμια, αλλά να μπορούν και να αποφυτούν με επιτυχία. Τώρα, για την ποιότητα, δύο στοιχεία θέλω να αναδείξω. Δύο στοιχεία. Διαχείριση και πρακτικές πρόσβασης. Ετήσεων. Κάποιες χώρες χρησιμοποιούν κεντρικοποιημένα συστήματα. Στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει το σύστημα Γιούκα, όπου όλοι οι φοιτητές ε, υποβάλλουν τις αιτήσει τους μέσω μιας κεντρικοποιημένης πύλης και στη συνέχεια αυτές οι αιτήσει ε, γίνονται αντικείμενο διαχείριση από τα επιμέρους πανεπιστήμια. Σε άλλες χώρες οι αιτήσει υποβάλλονται απευθείας στα πανεπιστήμια και υπάρχουν και κάποιες χώρες, ε, Γαλλία και Γερμανία είναι παραδείγματα, όπου υπάρχει ε, μια συνύπαρξη των δύο συστημάτων, δηλαδή και ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης και απευθείας το κεντρικό, το, κεντρικό σύστημα δηλαδή υποβολής αιτήσεων δεν υποκαθίσταται εντελώ, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία αποκέντρωση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προτίμηση από τη δική μας πλευρά στο ένα σύστημα ή στο άλλο, αλλά διαπιστώσαμε ότι αν κάποια χώρα θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον, τον δρόμο τη αποκέντρωση, τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πώ τα πανεπιστήμια ανταποκρίνονται για να χειριστούν όλε αυτέ τι διαδικασίε. Να διασφαλιστεί δηλαδή ότι το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων που ασχολείται με τη διαχείριση των αιτήσεων έχει τον κατάλληλη ε, προετοιμασία, εκπαίδευση, προκειμένου οι διαδικασίε αυτέ να διεκπεραιώνονται με ε, ποιοτικό, ε, υψηλά, με ποιοτικό τρόπο. Όσον αφορά το τι μα είπαν οι ενδιαφερόμενοι, τα, οι φορείς, οι οργανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να είναι τα πανεπιστήμια. Οι φορείς αυτοί θα ήθελαν επίσης ε, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Υπάρχει ήδη το, το δίκτυο Ανάντικ για την ε, αναγνώριση, την ισοτίμηση των ε, προσόντων, αλλά υπάρχει ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων προκτιών. Αναδεικνύεται αυτό το ζήτημα τουλάχιστον ως κάτι που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι είναι σημαντικό. Όσον αφορά τις πρακτικές πρόσβασης, ε, η χρονική συγκυρία επίσης έχει πολύ σημαντική, ε, είναι σημαντική και για τα πανεπιστήμια και για τους φοιτητές τα πανεπιστήμια που ε, διαχειρίζονται τα, τις αιτήσει λίγο πριν την έναρξη του, της σχολικής, της ακαδημαϊκής χρονιάς ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ιταλία και Γερμανία. Οι φοιτητές ε, συμπληρώνουν πάρα πολλές αιτήσει και αποφασίζουν τελευταίο, στο τελευταίο λεπτό σε ποιο πανεπιστήμιο τελικά θα πάνε. Σε περιπτώσεις που έχουν διάφορες προσφορές. Και αυτές οι καθυστερημένες αποφάσεις δημιουργούν προβλήματα στα πανεπιστήμια. Προφανώς. Στην Ιταλία υπάρχουν παρόμοια προβλήματα με τις εισαγωγικές εξετάσεις αν και υπήρχαν κάποιε αλλαγέ φέτο, αλλά οι εισαγωγικέ εξετάσει διεξάγονται λίγο πριν την, ε, την έναρξη της χρονιάς και έτσι οι φοιτητέ έχουν πολύ λίγο χρόνο να εξετάσουν ποιε είναι, είναι οι καλύτερε επιλογέ που έχουν στη διάθεσή του. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι οι κυβερνήσει μπορεί να εξετάσουν ε, το ενδεχόμενο να διενεργείται όλη αυτή η διαδικασία επιλογή νωρίτερα και όχι το Σεπτέμβριο. Just before... Και αυτό θα ήταν ακριβώς ε, πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Και το τελευταίο σημείο για τη σημασία της πληροφορίας για τα πολλαπλά κριτήρια. Όσο περισσότερες πληροφορίες λαμβάνουν οι ετούντες και όσο περισσότερες πληροφορίες λαμβάνουν τα πανεπιστήμια, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα και για τους δύο και για τα πανεπιστήμια και για τους φοιτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο επιλεκτικό το σύστημα. Πληροφορίες μπορούν να δίνονται ως ε, τμήμα της ε, συνεργασίας ε, μεταξύ πανεπιστημίων και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα τεστ. Η κινητικότητα τώρα αυξάνεται αρκετά. Βλέπετε ότι άλλαξε το ποσοστό μεταξύ 2005 και 2011. Παρ' όλα αυτά, Έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες ε, για την κινητικότητα αυτών που κάνουν αίτηση πρώτη φορά. Δηλαδή ξέρουμε πολλά για την κινητικότητα φοιτών μέσω του προγράμματος Εράσμους. Ξέρουμε ότι έχουν μεταβεί στο εξωτερικό αρκετοί φοιτητέ, ε, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η αναλογία των φοιτητών που αφού έχουν ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κάποια χώρα αποφασίζουν να κάνουν αίτηση και να πάνε στο πανεπιστήμιο σε μια διαφορετική χώρα. Αυτό το στοιχείο, αυτά τα στοιχεία θα ήταν πολύ ενδιαφέροντα να το αποκτήσουμε. Επίσης, ε, είδαμε ότι υπάρχουν πολλές φορές ε, κάποια εμπόδια στην κινητικότητα, Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα μεταφοράς ή αν θέτουν κάποιες ποσοστώσεις τα κράτη για συγκεκριμένα πτυχία σε σχέση με το πόσο που φοιτητές δεκτούν. Επίσης, το κόστος για να κάνει κανείς αίτηση στο εξωτερικό μπορεί να είναι υψηλό σε ό,τι αφορά ε, το κόστος ε, της συναλλαγής, πώς θα κάνει μια αίτηση σε μια ξένη χώρα, καθώς και τα ίδια ε, τα τέλη για την υποβολή της αίτησης. Μπορεί αυτά να είναι υψηλότερα για τους ελλοδαπούς φοιτητές. Έτσι λοιπόν με δύο λόγια, αυτά είναι τα πορίσματα σε σχέση με τις τρεις κυρίες διαστάσεις της μελέτες Υπάρχουν πάρα πολλά στην έκθεση, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο θα ξαναδώσω το λόγο στον συνάδελφο για να δούμε ποιες είναι οι συστάσεις πολιτικής που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέξαμε. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις έχουμε δύο σε ένα από τα κράτη-μέλη, ένα για τα κράτη-μέλη και ένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, ε κάποιες που θέλουμε να αναφέρουμε, κάποιες προειδοποίησεις. Καταρχήν, το θέμα της εισόδου είναι πολύπλοκο, έχουμε πολλές διαστάσεις, πρέπει να καταβάλουμε τι είδους τεστ, τι εξετάσεις έχουμε και επίσης θα πρέπει να κατανοήσουμε το είδος των απαιτήσεων αυτές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να καταλάβουμε πώς θα συντονίσουμε αυτά τα συστήματα. Επίσης, η δεύτερη προβλήση είναι ότι ε, έχουμε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα σε όλη την Ευρώπη για το θέμα της εισόδου, δηλαδή πώς επιλέγονται οι φοιτητέ. Και το τρίτο, ότι επειδή είναι επικοινόμορφα τα εθνικά συστήματα, καθώς και η εκπαίδευση είναι συμπληρωματική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές ε, για ε, κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω. Αυτές οι συστάσεις θα αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Για να επανέλθω τώρα ε, στις συστάσεις, ε, τι λέμε για την ισότητα για τα κράτη-μέλη, Τίνουμε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν ε, το θέμα της ισότητας, της εισόδου, ε, να προσπαθήσουν να παρέχουν περισσότερο διαφανείς πληροφορίες για τα συστήματα εισόδου. Αυτό σημαίνει όταν αυξάνεται η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων ε, και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι μαθητέ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να σκεφτούν τι πτυχίο θα ήθελαν. Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε το δυναμικό των μαθητών να ολοκληρώσουν τη δευτεροβαθμία εκπαίδευση ε, παρά απλώ να το για να μπουν στη τριτοβαθμία υπόδευση. Σε πολλέ χώρε το να μπορεί απλώ κάποιο να έχει πρόσβαση στο πανεπιστήμιο θεωρείται κάτι καλό. Εμεί δεν θεωρούμε ότι ε, είναι ο κατάλληλο τρόπο να προχωρήσουμε και επίση πρέπει να αξιολογηθούν οι τρέχουσε πρακτικέ ω προ το εισόδου των φοιτητών, κυρίω σε ό,τι αφορά του μη παραδοσιακού ε, εκπαιδευμένου Με αυτού θεωρούμε βασικά τους μαθητές που δεν ακολουθούν ε, το, την πεπατημένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά πάνε στο πανεπιστήμιο άνθρωποι που μπορεί να δουλέψουν ε, μεταξύ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του πτυχίου τους ή να αντικαταστήσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εδώ βλέπουμε μία διαφορά της αρχής ε, της μάθησης και της αναγνώρισής της ε, στην Ιταλία. Παραδείγματος χάρη η αναγνώριση είναι δυνατή όμως οι ετούντες θα πρέπει να έχουν και ένα ε, πιστοποιητικό, ένα πολιτήριο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν και αυτό το θέμα για τους μη παραδοσιακούς εκπαιδευμένους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προς την ισότητα σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Αυτό που βλέπουμε και αυτό που περιέγραψε ο Νικόλο είναι ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι αρκετά προσαρμοσμένα στις μεταρρυθμίσεις ε, που ακολουθήθηκαν από τα πανεπιστήμια στα τέλη δεκαετία του 90. Έτσι λοιπόν θα πρέπει τα πανεπιστήμια να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή ε, στο να έχουν το κατάλληλο προσωπικό ε, για την γραμματεία και να τους ενημερώνουν για τις πρακτικές, να ενημερώνονται για τα προσόντα τους. Επίσης δεν πιστεύουμε ότι είναι λογικό σε κάποιες χώρες να ξεκινούν οι εγγραφές τον Ιούλιο και σε κάποια άλλα να ξεκινάνε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Και σε ό,τι αφορά το σύστημα, συνολικά θα πρέπει ε, τα κράτη-μέλη να έχουν συγκεκριμένες κατευθύνες γραμμές και πρότυπα, καθώς και διαφανείς διαδικασίες ε, στην περίπτωση που κάποιο ετών δεν είναι ικανοποιημένος από τη διαδικασία της εγγραφής για την κινητικότητα μας εξέπλησε εξακολουθούμε να έχουμε κάποιες εκθέσεις που μας οδηγούν στο να πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια. Ε, έχουμε την περίπτωση του Βελγίου, παραδείγματος χάρη, ε, για την ιατρική υπάρχει ένα ποσοστό 13%. Εμείς ε, δεν πιστεύουμε ότι είναι λογικό να έχουμε δυσκολίες σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων υπάρχουν κάποια στοιχεία διμερών δυσκολίων εκεί. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια σε σχέση με την κινητικότητα των φοιτητών, ε, κυρίως σε ό,τι αφορά την ε, ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, πρέπει να δοθούν περισσότερα στοιχεία για τα μοντέλα της κινητικότητας σε ό,τι αφορά τώρα τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέμε ότι και η κινητικότητα αλλά και η συνεργασία είναι δύο τομείς όπου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αν το επιθυμούν φυσικά. Όσοι χαράσουν την πολιτική όπως είστε εσύ θα μπορούσαν να διαλέξουν το βασικό σενάριο αλλά αυτό το βασικό σενάριο δεν είναι η κατάλληλη εναλλακτική. Ίσως αυτό που θα συνέβαινε εδώ είναι ότι θα είχαμε θέματα και στην ποιότητα και στην ισότητα και θα είχαμε εμπόδια στην κινητικότητα, θα είχαμε υψηλό κόστο συναλλαγών για όσου θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ε, για να κάνει κάποιο κάποια αίτηση ανάλογα με τη χώρα κοστίζει από 40 έω 200 ευρώ. Αν θέλει ένα φοιτητή λοιπόν να κάνει αίτηση σε, σε τρει χώρε θα μπορούσε να έχει κόστο 600 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να λύσει αυτά τα εμπόδια. Για την ειδικότητα αναφερόμαστε σε δύο λύσεις λοιπόν. Ίσως η πρώτη είναι μια πιο ήπια επιλογή και έχει να κάνει με το να βοηθήσει τους επαγγελματίε ε, στον τομέα των ε, ε, εισόδων να ανταλλάξουν βέλτιστε πρακτικέ. Πολλοί Επαγγελματίε, ε, θα ήθελαν μια τέτοια πλατφόρμα ευρωπαϊκή. Έτσι λοιπόν η ιδέα είναι πάνω κάτω ίδια με αυτό που συμβαίνει σε άλλε χώρε, Παραδείγματο χάρη οι Πολιτείε Πολιτείε έχει την Διεθνή Ένωση για να παρέχει συμβουλέ για την ε, είσοδο στο κολέγιο. Έτσι λοιπόν η ιδέα θα ήταν να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για να βοηθήσουμε τι επαγγελματίε, να ανταλλάσσουν πρακτικέ και να καταλαβαίνουν ποια είναι τα κριτήρια ποιότητα. Αυτό έχει εφαρμοστεί επιτυχώ σε άλλου τομεί της τρίτοβάθμια εκπαίδευση, ε, Έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μητρό ε, το οποίο λειτουργεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Υπάρχει και μία τρίτη επιλογή η οποία ε, είναι η εξή να υποστηρίξουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μία διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών αιτήσεων. Έχουμε κάποιες πλατφόρμες στην πλουτίωση της Standing Europe που δίνουν πληροφορίες ε, στους ετούντες που θέλουν να φοιτήσουν στο εξωτερικό. Όμως δεν υπάρχει καμία πλατφόρμα όπου μπορούν να στείλουν οι φοιτητέ μία αίτηση που θα μπορούσε να σταλεί σε πολλά πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι πρωτοβουλίες υπάρχουν σε, ειδικά σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη Υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο μια πλατφόρμα που λέγεται Unicas ε, που βοηθάει τους Βρετανούς και Αγγλανδούς φοιτητές ε, να κάνουν αίτηση μέχρι και σε οκτώ πανεπιστήμια και αυτή η πλατφόρμα συλλέγει μία αίτηση και την διαχειρίζεται και τη στέλνει εκ μέρους των φοιτητών. Νομίζω ότι θα ήταν δίκαιο όλοι οι φοιτητέ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφελούνται από μια τέτοια πλατφόρμα, γιατί μπορεί να είναι μεγάλο το κόστος ε, της υποβολής αίτησης για τους φοιτητές αν θέλουν ε, να κάνουν τις σε διάφορες χώρες. Δεύτερον, γιατί το κόστος αυτών των διαφορετικών αιτήσεων επίσης ε, είναι υψηλό για τους οργανισμούς εισόδου, γιατί πρέπει να κατανοήσουν τις διάφορες διαδικασίες σε όλη την Ευρώπη και υπάρχει ένα κόστος για τα πανεπιστήμια και τα τριτοβάθμια ιδρύματα γιατί δεν ξέρουν τα πανεπιστήμια αν θα εμφανιστούν τελικά οι φοιτητέ όταν κάνουν διεθνεί αιτήσει. Έτσι, η ιδέα αυτή τη πλατφόρμα θα ήταν να μειωθεί το κόστο τη συλλογή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Φυσικά, για τις επιλογές αυτές ε, θα πρέπει να έχουμε μία περαιτέρω ανάλυση ε, κόστους κόστους-οφέλους, ε, για να δούμε αν θα είχε νόημα να προτιμήσουμε τη μία ή την άλλη επιλογή. Όμως, τονίζοντας αυτές τις επιλογές, πρέπει να τις τονίσουμε και σε σχέση με όσα έχουμε στην εκθεσή μας για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε και θα είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε οποιαδήποτε συνεισφορά σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη που ζητήθηκε στην προηγούμενη θητεία από την Επιτροπή Πολιτισμού. Εσείς μας παρουσιάσετε μια πλήρη έκθεση και με πίνακες και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη να δοθεί μια συνέχεια στην έκθεσή μας για την διαδικασία της Μπολόνια. Γιατί τίθενται αυτά τα μεγάλα τρία ερωτήματα για την ποιότητα, την ισότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών που μας ε, επιτρέπουν την κινητικότητα των ε, φοιτητών σε σχέση με την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και οι τρόποι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Έχετε συγκρίνει κάποια μοντέλα και από τα κράτη-μέλη αλλά και από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι οι συστάσεις σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Έχουμε και τα θέματα του χρόνου, ξέρουμε ότι υπάρχουν φοιτητέ, παιδιά συγγνώμη, που θέλουν να γραφτούν ή να κάνουν αίτηση σε διάφορα πανεπιστήμια, αλλά διαφέρουν οι χρόνοι για την υποβολή των αιτήσεων. Επίση, κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι η σύνδεση μεταξύ πρόσβαση και ισότητα. Δεν έχουμε μόνο του κανόνε ισότητα, αλλά και άλλου παράγοντε. Επίση, αναφερθήκατε σε ένα θέμα που είναι το θέμα της ε, ε, μεταφοράς, ε, χάρη, κάποιων υποτροφιών, ε, δηλαδή δέχονται κάποιες υποτροφίες, είναι δικαιούχοι κάποιων υποτροφιών οι και μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μόνο στο δικό τους πανεπιστήμιο. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών και σε άλλα πανεπιστήμια. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα είναι η έλλειψη στοιχείων. Εμείς ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός, ε, αλλά ξέρουμε μόνο τα στοιχεία για το Εράσμους. Από ό,τι κατάλαβα δεν ξέρουμε τη διαφορά ε, μεταξύ αιτήσεων και απαντήσεων. Δηλαδή αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όταν μιλάμε για την ε, ταξινόμηση των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να δούμε πόσο ανοιχτά είναι τα πανεπιστημιά μας και αν θα ρίνουν την κινητικότητα και κάτι άλλο ενδιαφέρον που είπατε. Το λέω γιατί αυτό είναι μια ιδέα για τη συζήτησή μας. Είναι το θέμα της ε, δυνατότητας δημιουργίας μιας πλατφόρμας. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί η ιδέα μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας ε, που να μας επιτρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα και μια συνολική διαδικασία εγγραφής ε, είναι κάτι που λείπει και τελικά έχει επίπτωση και στα αποτελέσματα. Νομίζω ότι μας παρουσιάσατε μια προβληματική εικόνα κατά κάποιο τρόπο. Καλό είναι ότι έχει αυξηθεί η κινητικότητα από το 2005, αλλά δυστυχώς ακόμη δεν γνωρίζουμε ε, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Φαντάζομαι θα θέλουν το λόγο συνάδελφοι. Παρακαλώ, συνάδελφος Μόργαν. <clears throat> Καταρχήν, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Νομίζω ότι πράγματι η απέτηση και η ευκαιρία για μια συγκριτική ανάλυση είναι κάτι σημαντικό και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ήταν και πολύ περιορισμένος ο χρόνος Και φυσικά αυτά που θέλω να υπογραμμίσω αφορούν και κάποια θέματα που έθιξε εκεί πρόεδρος. Καταρχήν, η μελέτη συνέκρινε 7 χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση και κάποιε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση. Το δεύτερο θέμα που μου φαίνεται σημαντικό σε σχέση με τα θέματα της ισότητας, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να δοθεί προσοχή όχι μόνο στην πρόσβαση στα ιδρύματα, δηλαδή τη στιγμή της εισόδου, αλλά και ε, στο αν ε, επιτυγχάνεται ε, η ολοκλήρωση των σπουδών. Επομένως πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα προσανατολισμού που υπάρχει σε διάφορα πανεπιστήμια έτσι ώστε οι φοιτητές να ακολουθούν κατά τις πανεπιστικές σπουδές μία συγκεκριμένη μυθοδολογία. Με συγχωρείτε, διακόπτη πρόεδρο. Συγγνώμη που σα διακόπτε, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα με του διερμηνεί. Ε, νομίζω ότι είναι εδώ ακόμα για 5-6 λεπτά. Πέρασε η ώρα, 12.30 έχει περάσει. Έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα λοιπόν. Ή μετά από 5 λεπτά, όποιο θέλει θα συνεχίσει στα αγγλικά. Ή μπορούμε να στείλουμε γραπτές ερωτήσεις στους ερευνητές μας Σα ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η λύση, αλλά ολοκληρώνω την υπηρεσία στη διερμηνία σε πέντε λεπτά. Ε, Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Θα ήθελα όμως ε, να ξαναπώ ότι ε, πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη σημασία ε, σε ένα στοιχείο που δεν είναι δευτερεύον, ε, δηλαδή τι γίνεται με το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί κάποιες χώρες το απαιτούν, κάποιες άλλες όχι. Μια άλλη πτυχή. Έχουμε κάποια μαθήματα με συγκεκριμένο αριθμό σπουδαστών που δέχονται συγκεκριμένο ρυθμό. και ολομένω περισσότερο στην Ιταλία υπάρχουν πανεπιστήμια που λόγω της αυτονομίας δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να κάνουν κάποια μαθήματα ακόμη και πριν πάρουν το απολυτήριο για να δουν στη συνέχεια ποιες δεν θα τους ενδιαφέρουν να επιλέξουν. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εξεταστεί και στο γενικό πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτό είναι και στο θέμα της ποιότητας. Επίσης, αν και καταλαβαίνω ε, τις απαιτήσει που εντοπίσατε, δεν θα υποτιμούσα το θέμα της αυτονομίας των πανεπιστημίων, γιατί ε, τίθεται και ένα θέμα α, καινοτομίας και αριστείας εδώ. Και τέλος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε και ένα ε, πολύ σημαντικό επιχείρημα για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία και κινητικότητα των εργαζομένων. Σεβόμενοι τι διάφορες κατευθυντήριε γραμμές που μας αναφέρετε, νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν παριθμόν 2. Γιατί δεν θα ήθελα για να φτάσουμε στον αριθμό 3 ε, να περάσουν κάποια χρόνια και να ξεκινήσουμε από το 0. Ευχαριστώ, Συνάδελφο Σομπρόβα. Και αν τα καταφέρουμε και οι υπόλοιποι. Děkuji. Já budu velmi stručná, protože chci Ευχαριστώ πολύ. Για να υπάρξει και δυνατότητα και άλλοι να παρεύουν πολύ σύντομα, είναι σημαντικό πιστεύω η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εποπτεύσουν τι γίνεται και πώς λειτουργεί ο τομέας αυτός συμπεριλαμβάνοντας και το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν έξι διαφορετικές περιπτώσεις έχοντας έξι, νομίζω αυτό δεν επαρκεί για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διαφορετικά τα συστήματα. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θετικά αυτή τη μελέτη, πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική μελέτη. Να δούμε τι συμβαίνει με τα 28 κράτη-μέλη, να συγκρίνουμε και να συναγάγουμε τα συμπεράσματα. Αυτό δεν επιτυγχάνεται με το σημερινό σύστημα των σημερινών περιπτώσεων. Το τι γίνεται δηλαδή σε σχέση με το δεύτερο βάθμιο τομέα εκπαίδευση και τον τρίτο βάθμιο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό είναι σημαντικό για να υπάρχει η διασφάλιση της ισότητα και θα πρέπει αυτό να ενταχθεί. Θα ήθελα επίσης να συστήσω να γίνει συνολική εποπτεία ολοκληρωμένη εποπτεία δεν είναι έργο νομίζω του Ευρωκοινοβουλίου. Θα πρέπει σε επαφή και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Λιμπάτσκα, νομίζω ότι είναι δυνατόν να πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Έτσι να έχουμε και διερμηνία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή η έκθεση οπωσδήποτε. Όμως θα ήθελα, αν γίνεται, να συνεχιστεί το έργο αυτό, να δοθεί συνέχεια, γιατί κάποιες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται. Ιδιαίτερα χώρες που η δημοκρατία βρίσκεται σε φθήνουσα απορία και συρρυκνώνεται και η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Και το πρόβλημα των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της ε, εισδοχής ε, συμπεριλαμβάνει μόνο πολύ λίγα θεσμικά όργανα, ε, εκπαιδευτικά όργανα κύρους και τίθεται το θέμα, το οποίο είναι θεμελιώδες ε, ζήτημα. Αν δεν υπάρχουν όρια ή φραγμοί, αν δεν υπάρχουν επίπεδα εξέτασης ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος ή όχι ένας υποψήφιος, μπορεί αυτό να δημιουργήσει απογοήτευση και να δούμε αν αυτό μπορεί να είναι θετικό ή όχι. Αλλά εδώ συνδέεται και ένα δευτερογενές επίπεδο σε σχέση με τα επίπεδα και τη διαφορετική δημογραφική κατάσταση κάποιων χωρών και όλα αυτά αφορούν την κινητικότητα και όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο. Και επίσης κάτι το οποίο βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ο βαθμός που ε, στο μέτρο του οποίου επηρεάζεται η ποιότητα μέσω αυτών των διαδικασιών. Πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε τη μελέτη ώστε να συμπεριληφθεί και αυτό το στοιχείο, λαμβάνοντας όσο το δυνατόν ευρύτερη η πληροφόρηση τι γίνεται σε σχέση με τις διάφορες χώρες μας. Φυσικά είναι αμφίδρομη η πορεία των πληροφοριών. Τι μπορεί να αναμένει ένας υποψήφιος από ένα εκπαιδευτικό όργανο σε σχέση με την αίτηση να γίνει δεκτός αυτό. Δεν είναι μόνο η έλλειψη γνώσεων πολλές φορές φραγμός, αλλά και η έλλειψη στοιχείων για να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των οργάνων. Και ένα τελικό ερώτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο όμως όταν έρχεται η ώρα να απαντηθεί. Θα πρέπει να υπάρχει αυτονομία των θεσμικών οργάνων, των εκπαιδευτικών οργάνων, να μπορούν εκείνα να ελέγχουν το σύστημα αποδοχής και εισδοχής υποψηφίων. Ευχαριστώ πολύ τους Δερμηνείς και μπορούμε να συνεχίσουμε στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Εδώ θα στημαρτήσουν οι υπηρεσίες ε, διερμηνίας. Γεια σας από εμά και λέει αν συμφωνείτε η Πρόεδρος να συνεχίσουμε στα αγγλικά στα γαλλικά και το λόγο έχει ο κύριος Κώστερ. Thank you for your presentation. It was very interesting and I think you have made clear that we need more findings and this is very important. I want to focus on the theme social inequality. I